Καλημέρα σε όλους, ευχές πολλές ε, για τα Χριστούγεννα και το καλό, τον καινούριο χρόνο. Έχουμε τα 10 και 11, τα οποία ε, θα αλλάξουν θέση, θα αντιστραφούν ε, και αν δεν έχετε ε, καμία αντίρρηση, τότε ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε την μέση διάταξη. Ε, γνωρίζετε πώς έχουν τα πράγματα. Έχετε όλες τις, ε, όλα τα σχετικά έγγραφα για την ε, επίσκεψη της αντιπροσωπείας την οποία είχαμε συζητήσει. 15 Ιανουαρίου, Δευτέρα, στις 7.30 ε, το απόγευμα θα κάνουμε μία έκτακτη συνεδρίαση των συντονιστών που όμως θα είναι ανοιχτή σε όλους τους συναδέλφους έτσι ώστε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Θα συζητήσουμε και τα θέματα θέματα τα οποία σχετίζονται με την διάσκεψη κορυφής ε, για την κλιματική αλλαγή, τη βιοπικιλότητα κτλ. Ε, και την κυκλική οικονομία. Στις 25 ε, θα έχουμε, Ιανουαρίου πάντα, θα έχουμε επίσης μια συνεδρίαση, αλλά ε, θα κάνουμε μόνο το απόγευμα συνεδρίαση ενώ θα ακυρωθεί η απογευματινή. Ε, όσον αφορά αλλαγέ στην γραμματεία μας ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον διοικητικό ε, που έρχεται από τη γραμματεία της ΣΥΜΚΟ και θα είναι μαζί μας επισήμως και από την 21η Ιανουαρίου. Επίσης να σας πω ότι θα έχουμε διαρμηνία ε, σε όλες τις γλώσσες όπως πάντα και ως ήθιστε. Είχαμε και μια συνεδρίαση των συντονιστών τον Δεκέμβριο. Ε, οι συστάσεις οι οποίες έχουν από αυτήν απορρεύσει έχουν ήδη ε, κυκλοφορήσει και αν δεν υπάρξουν σχόλια τότε ε, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Επίσης, ε, εάν μέχρι το τέλος ε, της συνεδρίασης ε, δεν έχουμε λάβει σχόλια για τις προηγούμενες συνεδριάσεις μας, θα θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά τους έχουν εγκριθεί. Τώρα θα περάσουμε στο πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. σχετικά με τον κανόνα 106. σε σχέση με επικαλύψεις οι οποίες έρχονται ε, σε επαφή με τα τρόφιμα. Θα ξεκινήσουμε όσοι ήθιστε δίνοντας το λόγο στον κύριο Χάουσλινγκ, στον ε, εισηγητή μας δηλαδή. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι ακόμα τώρα μπορούμε να ευχόμαστε καλή χρονιά, αλλά ξεκινάμε τη χρονιά με πολύ σοβαρή δουλειά και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ε, σχετικά με το κατά πόσον αυτά που κάνει η Κομισιόν σχετικά με, το, με την βιφενόλη Α ε, είναι η καλύτερη λύση και είναι κάτι ε, συνεκτικό με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προχωρήσει παραπέρα και επομένως να απαγορεύσει πλήρως την ουσία αυτή ε, και μάλιστα να το κάνει γρήγορα, πρέπει να ενεργήσει γρήγορα μια και πρόκειται για ε, ουσίες οι οποίες έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι σαφές ότι πρόκειται για ενδοκρινικό διαταράκτη, το γνωρίζουμε πλέον αυτό ε, είναι μια ουσία η οποία δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην ενδοκρινική λειτουργία ε, και στα ζώα και στους ε, ανθρώπους. Ε, είναι γνωστό αυτό σύμφωνα και με την έρευνα και την επιστημονική βιβλιογραφία. Δημιουργούνται προβλήματα στο κυκλοφορικό, δημιουργούνται προβλήματα γονιμότητας και επομένως είναι σαφές ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Και η μόνη λογική λύση είναι εν τέλει η απαγόρευση. Όμως διαπιστώνουμε ότι η Κομισιόν έχει άλλη άποψη. Έχουν γίνει κάποιες απαγορεύσεις ε, για τα μπιμπερόν, για τα ε, μπουκάλια για τα μωρά και τα πλαστικά ε, ποτήρια, αλλά και είναι καλό γιατί τα νεογνά και τα βρέφη προστατεύονται, αλλά υπάρχουν και τα μικρά παιδιά. υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. τι, τα μικρά παιδιά δεν πίνουν, ας πούμε, από πιο μεγάλα ποτήρια.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 ε, είναι γεγονός ότι ε, υπάρχει ε, και συσσόρευση ουσιών γιατί δεν έρχεται σε επαφή με τη δυσφενόλη μονάχα το, ο άνθρωπος αλλά και με ένα σωρό άλλες ουσίες οι οποίες είναι επιβαρυντικές και οι οποίες όταν σωρεύονται στον οργανισμό μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λέω λοιπόν ότι η μόνη λογική λύση είναι η κατάργηση και δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό με τον με, με, πανικό, θα πρέπει να δούμε αν εμείς ως Κοινοβούλιο ε, μπορούμε ε, να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα ε, από ό,τι είχαμε κάνει μέχρι τώρα. γιατί ας πούμε το είχαμε κάνει για τα υλικά γενικότερα και τις ουσίες που έρχονται σε επαφή ε, με τα τρόφιμα και σε εκείνη τη διαδικασία είχαμε πει ότι και ε, η δυσφενόλη θα πρέπει ε, να καταργηθεί. Η Γαλλία ας πούμε ήδη εφαρμόζει πλήρη απαγόρευση. Επομένως, Επομένως, είναι γεγονός ότι υπάρχουν 73 ουσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι γεγονός επίσης ότι κάποιες ουσίες ή κάποια υλικά ε, κοστίζουν περισσότερο από άλλες. Αλλά είναι γεγονός ότι εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν. Και γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτές τις ε, εναλλακτικέ λύσεις και να επιμένουμε πεισματικά στη χρήση της δυσφενόλης α. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να, ε, ε, ε, να μην επηρεαστούμε από την απόφαση της Κομισιόν και να ζητήσουμε την πλήρη απαγόρευση. Αυτό που προτείνει η Κομισιόν δεν είναι επαρκές και εμείς θέλουμε και πρέπει να πάμε παραπέρα. Και πιστεύω μάλιστα ότι θα πρέπει να γρηγορήσουμε. Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο γιατί πιστεύω ότι ε, και από πολιτικής απόψεως θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν εδώ. Το ζήτημα δεν είναι ποσοτικό, ε, έχει και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Και πόσες άλλες μελέτες επιτέλους χρειαζόμαστε έτσι ώστε να αποδείξουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος. Πρέπει πραγματικά να προστατέψουμε και το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε πιο σύντομοι γιατί δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Επόμενος ε, είναι ο κύριος ε, Μπαλάς Ε, που είναι συνεισηγητής. Εγώ στηρίζω αυτή την ένσταση γιατί, γιατί είναι λίγο, δεν στέκουν αυτά που λέει η Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει ότι υπάρχει πρόοδος και άρα θα στοχεύσουμε καλύτερα στην απαγόρευση της δυσφενόλης α, κυρίως για τα νεογνά. Αλλά ταυτόχρονα, εάν επιτρέπουμε τη δυσφενόλη α για τις εγγύες μητέρες ή για τα μικρά παιδιά, ε, δεν ρυθμίζεται το πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν εδώ μεγάλο πρόβλημα. Κάτι που είναι ακόμα πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου είναι το γεγονός ότι η Κομισιόν λέει θα μειώσουμε το κατόφλι και άρα θα παγορεύσουμε να υπάρχει περισσότερη δυσφενόλη α, θα βάλουμε συγκεκριμένα όριο δόσης. Το θέμα όμως είναι ότι οι ενδοκρινικοί διαταράχτες δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει κατόφλι. Σε πολύ μικρές δόσεις μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις και μάλιστα πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις από ότι με πιο, πιο μαζική ε, πιο μεγάλη δόση, δηλαδή εφέ κοκτέιλ σε συνδυασμό με άλλες ουσίες. Το γεγονός λοιπόν ότι μειώνεται το κατόφλι δεν αλλάζει και πολλά στην επικινδυνότητα αυτής της ουσίας της φαινόλης α. Δεύτερο, ε, τρίτο στοιχείο γιατί μας το προτείνει σήμερα η Κομισιόν αυτό, γιατί βασίζεται σε μια επιστημονική εκτίμηση της ΕΦΣΑ, της ε, υγειονομικής μας αρχής. Όμως η ίδια η αυτή αρχή αναγνωρίζει πως αυτή η μελέτη έχει πλέον ε, ε, ξεπεραστεί και μάλιστα έχει ξεκινήσει η διαδικασία για εκπόνηση νέας μελέτης που μάλιστα βρίσκεται στη φάση της δημόσιας διαβούλευση και αναμένεται να ολοκληρωθεί για το 2018. Άρα λοιπόν μας εντυπωσιάζει που βλέπουμε την Κομισιόν να, λαμβάνει τέτοιες, ε, να κάνει τέτοιες προτάσεις ε, για ένα δόγμα επιστημονικό το οποίο η ίδια το οποίο η ίδια η αρχή που το εξέδωσε το αμφισβήτη Υπάρχει λοιπόν μια, ένα πρόβλημα διαδικαστικό ε, πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο η Επιτροπή Περιβάλλοντος που εμείς είμαστε αυτοί, εμείς είμαστε αυτοί, ε, πρέπει να λάβουμε οπωσδήποτε θέση για το γεγονός ότι η Κομισιόν πρέπει να είναι λογική και να έχει σαν στόχο την πλήρη απαγόρευση των ενδοκρινικών διαταρακτών όταν έχουμε βρει την λύση αλλά και πιο συγκεκριμένα της δυσφενόλες α, γιατί ήδη ε, ισχύει σε κάποια ε, κράτη, ακόμα και αν δεν έχουμε βρει την εναλλακτική ακόμα λύση. Πώς λοιπόν η Κομισιόν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρίς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ε σας εύχομαι καταρχάς ε, καλή χρονιά και εγώ έχω συνυπογράψει την έσταση που κατέθεσε ο συνάδελφος Όσλινγκ για τη δυσφενόλη Α. Το είπαμε νομίζω αρκούντος ότι η Κομισιόν δεν προχωρά αρκετά μακριά για το σύνολο του θέματος των ενδοκρινικών διαταρακτών. Δεν θα επανέλθω στα φάσεις των τελευταίων μηνών, ούτε στην ιστορία των κριτηρίων, ούτε και στο θέμα συγκεκριμένα της δυσφαινόλης γιατί ο κύριος Χόσλινγκ το ανέλησε επαρκώς. Ε, ε, η Κομισιόν μας λέει ότι προτείνει για την αρχή της προφύλαξης γιατί μειώνει το κατά 10 φορέ επί 10 φορές σε όλες τις συσκευασίες, ε, ε, ε, τις πλαστικές συσκευασίες και καταργεί την δυσφενόλη τελείως για τα νεογνά και τα μωρά μέχρι τριών ετών, αλλά υπάρχουν και οι αγγείς γυναίκες, τα παιδιά άνω των τριών ετών, οι θυλάζουσες μητέρες που δεν τους έχουμε αναφέρει ακόμα. Πολλές μελέτες δείχνουν πόσο ευαίσθητες είναι οι αγγείς γυναίκες σε ρήπους τέτοιους οργανικούς. Ε, το έχουμε αυτό αναφέρει στα εκτιμώντας νη και πι, εν και πε. Άρα λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν μου φαίνεται πως είναι ένας τρόπος να νομιμοποιήσει και να αποκαταστήσει τη χρήση μιας χημικής ουσίας που όλο ένα και ε, περισσότερο είναι αντικείμενο ε, προσοχή. Η Κομισιόν φαίνεται να έχει λοιπόν ε, κολλήσει στο χρόνο ε, έχει, το 2015 σε εκείνη τη μελέτη που λέει ότι το δυσφενόλη α δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει έκτοτε. Αυτά τα συμπεράσματα είναι ξεπερασμένα, εκπίπτουν γιατί ε, τον Ιούνιο του 2017 ελήφθη απόφαση από τους εμπειρογνώμονες ε, της, των ειδικών για τα χημικές ουσίες που λένε ότι είναι εξαιρετικά ψηλή επικίνδυνη μάλιστα η δυσφενόλη α, διότι είναι ενδοκρινικός διαταράχτης. Αυτά στο πλαίσιο των αναλύσεων του ΡΙΤΣ Δεν υπάρχει πλέον καμία αντίφαση δηλαδή, δεν ε, συνεχίζεται συζήτηση όπως για το γλυφοσάτι. Εδώ η Κομισιόν θα πρέπει να ακολουθήσει τη γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων η μόνη, λοιπόν, το μόνο συμπέρασμα είναι αυτό που οδηγεί στην απαγόρευση σε κάθε συσκευασία τροφίμων. Ε, Υπήρξαν σχετικές αποφάσεις και μελέτες και στη ΣΥΠΑ. Είδαμε, ε, είδαν εκεί από το 2006 ότι η δυσφενόλη Α έχει επιρροή ακόμα και σε χαμηλές δόσεις ε, στα δοκιμές ε, Γι' αυτό και καταλήγω στο εξή. Οι πολίτε ε, έχουν βαρεθεί αυτά τα πηγενέλα, τα δύο βήματα μπροστά και τρία πίσω. Ε, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να επιμείνουμε εδώ και να επιβεβαιώσουμε την ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλειά μα τον Οκτώβριο του 2016 υπέρ τη απαγόρευση αυτή. Γιατί είναι πραγματικά τρελό το να κάνουμε πίσω σε σχέση με αυτό που έχουμε ήδη ψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ.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 ότι αυτά που αποφάσισαν, αποφάσισε η Επιτροπή είναι λογικά. Ιδιαιτέρως δε, διότι η Επιτροπή ζήτησε από την ΕΦΣΑ να ασχοληθεί με το θέμα και ε, να διεξάγει μελέτες. Ε, και η ΕΦΣΑ πάντοτε λαμβάνει υπόψη της και άλλες μελέτες που έρχονται ας πούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι ε, ε, εκεί πρέπει να βασιστούμε. Είναι γεγονός ότι κάποιες χώρες έχουν πιο αυστηρά όρια και αργότερα βέβαια μπορούμε να δούμε και εμείς εάν είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε παραπάνω και επομένως δεν δέχεται την αντίρρηση αυτή το ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, έχω και μία επιπλέον ερώτηση προς την ε, Κομισιόν. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ποιες ε, είναι οι επιπτώσεις ε, αυτού του κανονισμού στην γαλλική απαγόρευση της δυσφενόλης. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, λέει η κυρία Σαλντεμόζε, ε, θέλω να πω το εξή ε, κάτι που ήταν προφανές και σαφές από την αρχή, δηλαδή ότι ε, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι απολύτως υπέρ της πλήρους κατάργησης και αυτής της ουσίας και κάποιων άλλων που δεν είναι της παρούσης. Είμαστε λοιπόν υπέρ πλήρους απαγόρευσης. Πιστεύουμε ότι εδώ μιλάμε για μια επικίνδυνη ουσία και επομένως είναι καλό να μένει μακριά από τα τρόφιμά μας και δεν πιστεύουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχωράει αρκετά μακριά. Πρέπει να είμαστε ε, και να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία, να είμαστε πιο ε, ε, να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία και επομένως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την αντίρρηση θα πρέπει να δώσουμε στους εαυτούς μας την ε, δυνατότητα ε, να ε, διεκδικήσουμε την απαγόρευση και όμως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορούμε να συζητήσουμε και να ζητήσουμε περαιτέρω ε, νομοθεσία. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί τώρα ε, να μην ε, μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε να κάνουμε παρόλα αυτά αποτελεί ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και επομένως δεν θα συμφωνήσουμε με την αντίρρηση αυτή γιατί πιστεύουμε ότι έστω και αυτό το μικρό βήμα είναι καλό ε, Αλλιώς θα κλείσουμε τελείως τις νομοθετικές δυνατότητες και πόρτες. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στο μέλλον. Όταν θα έχουμε την νέα επιτροπή μετά από, το, ε, από τις νέες ευρωπαϊκές ε, εκλογές, ίσως θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο γενικό σχέδιο και σχεδιασμό για όλους τους ε, ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες. Το σημαντικό σήμερα είναι να αφήσουμε πόρτες ανοιχτές, να κάνουμε το πρώτο βήμα έτσι ώστε να αρχίσουμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Και μπορούμε ε, να το κάνουμε το δεύτερο βήμα μετά από έξι μήνες. Επομένως εμείς θέλουμε να πάρουμε αυτό το μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. και αν η πρόταση περάσει θα πρέπει ε, να βεβαιωθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τακτικό χρονικά διαστήματα μας ενημερώνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε ε, να γνωρίζουμε την κατάσταση, πώς προχωράει η εφαρμογή στα κράτη-μέλη κτλ. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την αντίρρηση γιατί ε, ε, πιστεύουμε ότι ναι, τώρα είναι λιγότερο καλή η προστασία των παιδιών, ε, των βρεφών, αλλά ανοίγουμε μια καλή πόρτα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούλικεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους, λέει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει ένα σημείο με το οποίο μπορώ να συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Χόισλινγκ, δηλαδή ναι, συζητούμε ένα πολύ ε, σημαντικό και ενδιαφέρον ζήτημα. Όσον αφορά τα, ε, τα όσα προτείνει η Κομισιόν, ε, πιστεύουμε ότι είναι ουσιώδη και μπορούν σημαντικά να βελτιώσουν την παρούσα κατάσταση και μάλιστα από τώρα και επομένως πολύ γρήγορα άματη εφαρμογή. Ε, θα ήθελα να θυμίσω τα σημεία τα οποία είναι σημαντικά σε αυτό το νομοθέτημα. Καθορίζει ένα πολύ πιο, μια πολύ πιο χαμηλή υποχρεωτική τιμή για την ε, δυσφενόλη. Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται είναι Ε, από το 0,6 πήγαμε στο 0,005 και επομένως έχουμε μία μείωση 10 ε, ε, φορές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό έλαβε υπόψη της η Κομισιόν. Επιπλέον έχουμε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, πράγμα επίσης πολύ σημαντικό και εκτός από τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουμε πλέον και την χρήση δυσφενόλης ε, σε επιχρήσματα, σε επικαλύψεις ε, σκευών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πράγμα που μειώνει σημαντικά την έκθεση στην βυσενόλη α. Επίσης και τρίτον η Κομισιόν έλαβε υπόψη τις διάφορες διατάξεις που ήδη ισχύουν ε, ε, σε ορισμένες χώρες ε, και έλαβε υπόψη ας πούμε την περίπτωση της Γαλλίας και έλαβε υπόψη την αρχή της πρόληψης και την εφαρμόζει την ρήτρα πρόληψης σε αυτές τις περιπτώσεις Επίσης η Κομισιόν ε, γνωρίζει βεβαίως όλη την εργασία η οποία έχει ξεκινήσει από το 2015 ε, και στην ε, γενικό, στο γενικότερο θέμα των χημικών ε, ουσιών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δυσφενόλη, έλαβε υπόψη την εργασία της ΕΦΣΑ, διότι ε, ο οργανισμός αυτός έχει μελετήσει διεξοδικά την επίδραση του στοιχείου αυτού στον οργανισμό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ΕΦΣΑ επίσης μελέτησε ε, την ε, ε, έκθεση των ανθρώπων στην δυσφενόλη και τα αποτελέσματα που θα μπορούσε αυτή να έχει. Η ΕΦΣΑ βεβαίως έλεβε υπόψη και την δυσφενόλη ως ορμονικό διαταράκτη Όσον αφορά κάποιους από τους προβληματισμούς που αναφέρονται στο ψήφισμα, η Κομισιόν γνωρίζει ότι μπορεί στο ανακυκλωμένο χαρτί να βρεθούν ίχνη δυσφενόλης α, ε, αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση ε, για ε, σκοπίμως προστιθέμενη ουσία στη διάρκεια της ανακύκλωσης ναι, μπορεί να υπάρξει μια ε, τέτοια έκκληση. Ε, ε, θα πρέπει να μελετήσουμε ξανά το θέμα αυτό όταν θα έχουν εφαρμοστεί όλες οι διατάξεις που αφορούν και την ανακύκλωση μέχρι το 2020. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η δράση η οποία έχει ήδη αναλυφθεί από ορισμένε χώρες μέλη και από την βιομηχανία. Η Γαλλία αναφέρθηκε προηγουμένως, αλλά μπορούμε να πούμε ότι και η Δανία και η Σουηδία και το Βέλγιο έχουν ε, σε εθνικό επίπεδο ορίσει περιορισμούς. Ε, αυτά τα στοιχεία ελήφθησαν υπόψη από την Κομισιόν στη σύνταξη του νομοθετήματος. Ε, γνωρίζομαι τις προσπάθειες της βιομηχανίας για αντικατάσταση της δυσφενόλη και λαμβάνουμε βεβαίως υπόψη και τις σχετικές απαγορεύσει των κρατών μελών. Υπάρχουν δυσκολίες συμπαραλαμβανομένης ας πούμε της έλλειψης ασφαλούς και επιβεβαιωμένης ε, εναλλακτικής ε, ουσίας. Ε, έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες αντικτύπου και σκοπιμότητας για εναλλακτικές ουσίες και όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη και στην προαναφερθήσα γαλλική απαγόρευση ε, γιατί ε, ε, αναφέρεται άλλωστε ότι ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα δοχεία τροφίμων αλλά και τα, οι τρόποι μεταφοράς ας πούμε μεγάλες δεξαμενές μέσω των οποίων γίνεται μεταφορά τροφίμων. Ε, ε, υπάρχει μια ερώτηση επίσης σχετικά με το κατά πόσον η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη τον αντίκτυπο ε, επί του νομοθετήματος των γαλλικών μέτρων. Σας είπα και προηγουμένως ότι εν τέλει δεν πρόκειται για πλήρη απαγόρευση ούτε και στην Γαλλία. Οπωσδήποτε θα έρθουμε όμως ως Κομισιόν σε επαφή με τις γαλλικές αρχές έτσι ώστε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει κάποια επικάλυψη και ενδεχομένως να ζητήσουμε από τη Γαλλία να αναθεωρήσει κάποια μέτρα και εν πάση περιπτώσει κατά αυτή την έννοια θα υπάρξει μια ε, μέτρηση και μελέτη της ε, διαφοράς που ενδεχομένως θα προκύψει. Αυτό που θέλουμε ε, να υπογραμμίσουμε είναι το εξής. Εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Ξέρετε ότι η Κομισιόν έχει ζητήσει από την ΕΦΣΑ να ξεκινήσει μια πλήρη αναθεώρηση και μελέτη της της φερνόλη α. Και ε, αναμένουμε ε, ε, ε, ε, το αποτέλεσμα αυτής της πλήρους επανεξέτασης από βάση της ΕΦΣΑ περί τα τέλη του 2019. Εν τω μεταξύ δηλαδή εργάζεται η ΕΦΣΑ επί του θέματος αυτού και η Κομισιόν συνεχίζει να ασχολείται με το θέμα και βεβαίως η υπό την αίρεση των αποτελεσμάτων που θα τις κοινοποιήσει η ΕΦΣΑ ενδεχομένως θα αλλάξει και την στάση της. Αυτά όσον αφορά τους στόχους του κανονισμού μεταξύ των οποίων και ε, κυρίως η προστασία της ε, ανθρώπινης υγείας και πρέπει να πω ότι ε, το μέτρο ως έχει, έχει ήδη υποστηριχθεί από 27 χώρες από τις 28 και ε, πιστεύουμε ότι με την πλήρη απόρριψη αυτού του νομοθετήματος αυτή τη στιγμή εν τέλει ε, θα ε, ζημιώσουμε την ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση περί αυτής της ένστασης. Θα ψηφίσουμε αργότερα. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Πού είναι οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Ετοιμάστε τις κάρτες σας παρακαλώ. Two objections. the other one is the early non-objection, the one on ETS aviation Brexit. Okay, is anyone, everyone seated? Yeah.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 την ένσταση για την δυσφενόλη α ηλεκτρονικά. Οπότε άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Δεν βλέπω Okay, everyone voted, then vote is closed. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. And the last vote. Yes. yes. Is on a, a draft recommendation. Επόμενη ψηφοφορία, σχέδιο σύστασης για υποβολή ένσταση για το σχέδιο ε, κανονισμού ε, της Κομισιόν που θεσπίζει Μητρό Ένωσης. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Αγκρίνεται. Mm. Τέλος των ψηφοφοριών. Και επόμενο μας θέμα είναι σε δύο λεπτά με τον Επίτροπο Στυλιανίδη. Σας καλώ να μείνετε για την ανταλλαγή απόψεων. Σε ένα-δύο λεπτά είναι εδώ.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

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε πάλι και ε, καλωσορίζω και εκ μέρου σας βεβαίως τον Επίτροπο κ. Στυλιανίδη. Η σημερινή του επίσκεψη έχει σχέση και με την δημοσίευση της προτάσεως για την τροποποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. Το θέμα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και βέβαια και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, συμβαίνουν πολλές θεομηνίες και άλλες ε, φυσικές καταστροφές. Είναι σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί για την αντιμετώπιση τους. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θα δώσω μέσα το λόγο στον Επίτροπο και μετά έχω ήδη σημειώσει ορισμένα ονόματα στην λίστα για να μπορέσουν οι ευρωβουλευτές να θέσουν ερωτήσεις. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Αλλά χωρίς μικρόφωνο. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα καλή χρονιά και τις καλύτερες ευχές μου για σας και τις οικογένειές σας. Όπως είπε η πρόεδρό σας, θα συζητήσουμε τις προτάσεις μας για την διάσωση. Έχω ακούσει ορισμένους από εσά ξεχωριστά. Αυτή τη φορά έρχομαι στην Επιτροπή σας και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών, ευρωπαϊκών μηχανισμών διάσωσης και χαίρομαι που επιληφθήκατε με ταχύτητα των προτάσεών μας. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο. Η κοινή μας προτεραιότητα είναι να ενισχύσουμε τον μηχανισμό όσο γίνεται γρηγορότερα για να μπορέσουμε να προλάβουμε, να προετοιμαστούμε και να ανταποκριθούμε στις καταστροφές. Να σώσουμε ζωές πρώτα-πρώτα και περιουσίες των Ευρωπαίων πολιτών προς το συμφέρον των πολιτών μας και βέβαια να προστατεύσουμε το περιβάλλον διότι δυστυχώς η επόμενη θεομηνία περιμένει για να ξεσπάσει σήμερα γνωρίζετε και καλύτερα από μένα διότι ως μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχετε σχετική γνώση, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτά δεν είναι fake news. Και επιμένω επ' αυτού. Όλο και συχνότερες και εντονότερες πλημμύρες θύελες, πυρκαγιές δασών, και μια φορά ταυτόχρονα σε πολλές χώρες και γνωρίζουμε ότι βεβαίως οι θεομηνίες δεν γνωρίζουν ούτε κρατικά σύνορα. Πρώτα, οι φυσικές καταστροφές βεβαίως πλήττουν τους ανθρώπους, τις περιουσίες τους, το βιός τους, την υγεία και την ασφάλειά τους. Το ίδιο προβλήματα αντιμετωπίζουν κάποιοι ζωτικοί οικονομικοί τομείς από την Αλία μέχρι τη Δασοκομεία και τη Γεωργία. Δεύτερο, οι φυσικές καταστροφές πλήττουν το περιβάλλον και βεβαίως ταυτόχρονα και τη βιοπικιλότητα. Τα οικοσυστήματα είναι ευάλωτα σε αυτές τις κρίσιμες αλλαγές. Φυτικά και ζωικά είδη κάνουν αγώνα για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και τρίτο είδαμε πολλές φορές το αποτέλεσμα αυτό των φυσικών καταστροφών που είναι ότι καταστρέφει και πολιτιστική κληρονομιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λόγω των βροχοπτώσεων, λόγω και της ε, αύξησης του επίπεδου των θαλασσών. Για όλους αυτούς τους λόγους οφείλω να επιμείνω ότι η κλιματική αλλαγή διόλου δεν είναι ψευδής ειδήσει. Είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς ε, πάει και να γίνει ο νέος κανόνας. Και κάθε ένας, όλοι οι παγκόσμιοι ηγέτες οφείλουν να αναγνωρίσουν τη σκληρή αυτή νέα πραγματικότητα. Και γι' αυτό ως Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στοχεύουμε ήδη και επιμένουμε στην απαράβατη τήρηση της Συμφωνίας του Παρισιού που είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την βαθιά αυτή αλλαγή που επέρχεται στις ζωές μας. Ουδής πρόκειται να τη γλιτώσει. Από το βορρά έως τον νότο, από τη δύση έως την ανατολή δεν υπάρχουν όπως είπα όρια. Είδαμε σήμερα το πρωί. Σε διάφορα κανάλια, το CNN, το BBC, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είδαμε σχετικά με τις καταστροφικές πλημμύρες στην Καλιφόρνια και στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δέστε τι γίνεται και εδώ στη δική μας Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τι έγινε δηλαδή στο 2017. Πραγματικά ήταν ένα δραματικό έτος από την άποψη αυτή. Με πυρκαγιές δασών στην Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, χωρίς προηγούμενο, ακόμα και στην Ιρλανδία, στο Μαυροβούνιο, στην Αλβανία, στην Τινησία. Γνωρίζετε ότι προδιετίας αντιμετωπίσαμε πυρκαγιές δασών στην Γρυλανδία. Κάτι το ε, απολύτως απροσδόκητο. Πυρκαγιές δασών στη Γρυλανδία. Ταυτόχρονα ο τυφώνας οφιλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα, βαρύτατες πλημμύρες, θανατηφόρες θύελες και στην Ελλάδα και στην ε, Γερμανία και αλλού. Θεομηνίες οι οποίες έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θυμάτων, βαρύτατες οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ή στατιστικές δείχνουν ότι οι ζημιές φτάνουν στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ 10 δισεκατομμύρια ευρώ ζημιές το 2016 στην Ευρώπη. Επομένως, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές γίνονται και πιο συχνές και πιο βαριές, πλήττουν όλο και περισσότερες χώρες μέλη και οι επιπτώσεις τους είναι πιο απρόβλεπτες ακόμη και προκαλούν κατεπίγουσες καταστάσεις που ξεπερνούν τους εθνικούς πόρους και τις εθνικές ικανότητες ακόμα και στις μεγάλες χώρες μέλη μας. Πρόσφατες φυσικές καταστροφές αποδείχνουν ότι οι φυστάμενοι προληπτικοί μηχανοί, μηχανισμοί συγγνώμη, και μέτρα δεν επαρκούν. Μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν όλοι ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο για μια Ευρώπη η οποία επιθυμεί να προστατεύει τους πολίτες της, τους πολίτες μας. Οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις δυνατότητές μας στις νέες πραγματικότητες, να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να ανταποκρινόμαστε και για να προλαμβάνουμε. Όπως είπε ο Ζωάν Κλοντ Ιούνκερ θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει κάτι παραπάνω από τα συλληπιτήριά της όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες θεομηνίες. Ο τρέχον μηχανισμός πολιτικής προστασίας επιτύχει πολλά πράγματα. Ως Επίτροπος Αρμόδιος για το μηχανισμό αυτό είμαι υπερήφανο για το υφιστάμενο σύστημα διότι είδα επιτόπου πολλά επιτεύγματα που οφείλονται στην ε, χρήση του μηχανισμού αυτού, της δομής αυτής. Η δομή αυτή, το παρόν σύστημα, βασίζεται σε οικειοθελείς συνεισφορές των χωρών μελών μας και είμαι βαθύτατα ευγνώμων σε όλες τις χώρες μέλη και σε όλες τις διοικήσεις που έδειξαν αλληλεγγύη προς άλλες χώρες σε περιόδους κατεπηγουσών καταστάσεων. Όμως, το οικειοθελές αυτό σύστημα έχει φτάσει πλέον στα όρια του. Λόγω των νέων και βαρύτερων επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής. Και διότι και το επαναλαμβάνω αυτό και διότι λέω αντιμετωπίζουμε πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα σε διαφορετικές χώρες. Το 2017 οι αιτήσει για βοήθεια παρέμειναν αναπάντητες. Μόνο 10 από τις 17 αιτήσει στη διάρκεια των πυρκαγιών δασών μπόρεσαν να απαντηθούν πλήρως. Καμιά φορά μπορέσαμε να δώσουμε βοήθεια πολύ αργότερα, μετά από την έκτακτη κατάσταση. Το είδα αυτό επιτόπου και ήταν μια οδυνηρή εμπειρία για μένα ως Ευρωπαίο αξιωματούχο. Στην διάρκεια των πυρκαγιών δασών στην Πορτογαλία, πέρσι τον Οκτώβριο, ακόμα και χώρες με ισχυρό ιστορικό αλληλεγγύης δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν διότι είχαν ήδη ξεπεραστεί οι ικανότητές τους από τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν στις ίδιες τους τις χώρες. Και από αυτή την οδυνηρή εμπειρία στην Πορτογαλία αντιληφθήκαμε ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη να αυξήσει την συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης των καταστροφών. Γι' αυτό το λόγο τον Νοέμβρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναβαθμίσει τον προληπτικό μηχανισμό και να δημιουργήσει την διάσωση, ρέσκιου. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους μου του Σώματος των Επιτρόπων, διότι μπορέσαμε να εγκρίνουμε τις προτάσεις αυτές ομόφωνα. Πολύ εξημών Γνωρίζετε ήδη τις προτάσεις αυτές, αλλά να μου επιτρέψετε να τονίσω κάτι που έχει κρίσιμη σημασία, διότι ήδη έχω ξεκινήσει σειρά επισκέψεων στις χώρες μέλη και συναντήσεων και θέλω να διευκρινίσω κάποια παρανόηση. Η διάσωση, rescue δηλαδή, δεν θα αντικαταστήσει τα όσα κάνουν οι χώρες μέλη. Δεν θα υποκαταστήσει. Η βασική ευθύνη για την αντιμετώπιση των θεομηνιών είναι και εξακολουθεί να είναι υπόθεση των χωρών μελών. Άρα η Rescue θα συμπληρώνει τις προσπάθειες των χωρών μελών όταν και όπου αυτό είναι αναγκαίο. Όταν και όπου οι εθνικές ικανότητες και πόροι δεν επαρκούν. Με άλλα λόγια, ο μηχανισμός Rescue θα είναι ένα δίχτυ ασφαλείας όταν θα αντιμετωπίζουμε εξαιρετικές καταστάσεις, εξαιρετικές έκτακτες καταστάσεις, να το πω καλύτερα έτσι, όπου δεν επαρκούν τα εθνικά μέσα. Πρόκειται δηλαδή για μια στην πράξη εφαρμογή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης όταν οι εθνικοί πόροι δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένη καταστάσεως. Σύντομα τώρα να σας εξηγήσω την πρόταση για τον μηχανισμό Rescue. Πρόκειται για δομή βασισμένη σε δύο πυλώνες οι οποίοι οι πυλώνες είναι ισορροπημένοι και αλληλοεξαρτώνται και γι' αυτό τονίζω ιδιαίτερα τον ισχυρό σύνδεσμο μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης γιατί και οι δύο αυτοί πυλώνες είναι το ίδιο σημαντικοί αλληλεγγύη και ευθύνη διότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η αλληλεγγύη οφείλει να ακολουθεί την ευθύνη. Είμαι απόλυτα πεπισμένος για την ορθότητα του επιχειρήματο αυτού και αυτό προέρχεται και από την εμπειρία σε αυτόν τον πολύ απαιτητικό τομέα. Πρώτος λοιπόν πυλώνας είναι ο Rescue. Με τον Rescue η Ένωσή μα, θα έχει δικές της ικανότητες να ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφέ με δικό της έλεγχο και διοίκηση στα τρία επίπεδα της πυραμιδικής δομής. Νομίζω ήδη τα έχουμε πει αυτά. Εκ παραλλήλου βέβαια θα αυξήσουμε τα οικονομικά κίνητρα για τις χώρες μέλη για να διαθέσουν ικανότητες που διαθέτουν και σε άλλες χώρες. Για να μπορούν δηλαδή να μεταφέρουν, να επιδιορθώνουν, να μεταφέρουν και να χρησιμοποιούν μηχανήματα και άλλα μέσα αλλού. Civil Protection Pool το λέμε αυτό και είναι ένα είδος αναβάθμισης του ε, υφιστάμενου συστήματος το οποίο είναι όπως είπα σε βάση εθελοντική. Να έρθω τώρα στο δεύτερο πυλώνα των προτάσεων πρόληψη και προπαρασκευή. Αυτή είναι και η προσωπική μου μανία να το πω έτσι. Χωρίς πρόληψη και προετοιμασία δεν πάμε πουθενά. Χρειαζόμαστε προσεκτικά σχεδιασμένη και συντονισμένη πρόληψη εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σε βάθος τις φυσικές καταστροφές. Παράδειγμα, χθες μόλις οι ερευνητές σε Ινστιτούτο Ερευνητικό Ινστιτούτο στη Γερμανία πραγματικά πολύ φημισμένο δημοσίευσαν μελέτη για την αύξηση του κινδύνου πλημμυρών λόγω της αλλαγής του pattern των βροχοπτώσεων. Και δείχνει η μελέτη αυτή ότι χρειάζονται και παγκοσμίω αλλά και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και ιδίω στην κεντρική Ευρώπη νέοι σχεδιασμοί για την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Προσαρμογή, επομένω, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, γιατί η προσαρμογή σημαίνει στην πραγματικότητα πρόληψη και προετοιμασία. Σήμερα έχουμε δεν έχουμε μάλλον κανένα ρόλο ως ευρωπαϊκοί θεσμοί στην πρόληψη και προετοιμασία. Ορισμένες φορές δεν γνωρίζουμε καν ούτε αν οι χώρες μέλη μας το κάνουν αυτό. Θέλουμε όμως οι χώρες μέλη να έχουν σχεδιασμό αξιολόγηση του κινδύνου. Εύκαμπτο σχεδιασμό, προσαρμοσμένο σχεδιασμό για την αξιολόγηση των κινδύνων. Και θα στηρίξουμε τι προσπάθειε των χωρών μελών προ την κατεύθυνση αυτή. Θα τι βοηθήσουμε επίση να φτιάξουν μια κοινή κουλτούρα, μια κοινή νοοτροπία για, την, για το σχεδιασμό αυτό. Θα προσφέρουμε τεχνογνωσία για να φτιαχτεί ένα δίκτυο, ενωσιακό δίκτυο για την πρόληψη. Το ίδιο και αυτό είναι το άλλο μέρος της πρότασής μας για πρόληψη και προετοιμασία τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μπορούν να προσφέρουν σημαντική στήριξη, χρηματοδοτική στήριξη στις χώρες μέλη για τον σχεδιασμό πρόληψης και προετοιμασίας. Όλη η εμπειρία μας αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε τον συντονισμό αυτό μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων έτσι ώστε να δώσουμε στις χώρες μέλη μας περισσότερα κίνητρα για να κινητοποιηθούν περισσότερο για την πρόληψη και προετοιμασία. Και βέβαια οι χώρες μέλη θα πρέπει να υποστηριχθούν και μέσω όλων των σχετικών ενωσιακών πολιτικών περιβάλλοντος, κλίματος, υγείας και έρευνας ως παραδείγματα. Τέλος, αλλά ουχή λιγότερο σημαντικό. Ο μηχανισμός Rescue αναφέρεται σε οικονομίες κλίμακος και είναι ο ορισμός των οικονομικών κλίμακος και στην ανταπόκριση αλλά και για την προετοιμασία. Ο Rescue λοιπόν αναφέρεται στην μέγιστη αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη γραφειοκρατία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Rescue αποδεικνύει την δέσμευσή μας για να αυξήσουμε την στήριξη της Ένωσης προς τους πολίτες όταν θεομηνίες, φυσικές καταστροφές απειλούν τις, ζωής, τις ζωές τους, τις περιουσίες τους, το περιβάλλον τους. Πολλοί από εσά έχετε εκφράσει ενδιαφέρον και υποστήριξη και ευχαριστώ βεβαίω και για την θερμή υποδοχή που επιφυλάξατε τις προτάσεις αυτές στο Στρασβούργο τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Και βεβαίως χρειάζεται ταχεία εκκίνηση της νομοθετικής διαδικασίας. Δεν είναι μυστικό ότι η επόμενη φυσική καταστροφή θα χτυπήσει ανα πάσα στιγμή. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα και γι' αυτό είναι κρίσιμο να έχουμε τον μηχανισμό μας έτοιμο να λειτουργήσει το δυνατόν συντομότερο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την ομιλία μου και πολύ ευχαρίστως ακούω ερωτήσεις, σχόλια προτάσεις και πιστεύω απολύτως ότι όλοι συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες αυτές αλλά και την άποψη ότι το υφιστάμενο σύστημα πρέπει να αναβαθμιστεί για να μπορέσει να αρθεί στο ύψος της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μιλήσατε για έκτακτες καταστάσεις, μιλήσατε για την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού. Αυτό μας απασχολεί και μας εντόνως. Δεσμεύεται η Επιτροπή μας να εργαστεί με ταχύτητα για να προσπαθήσει να είναι έτοιμος ο μηχανισμός αυτός για το επόμενο καλοκαίρι. για καλύτερη προετοιμασία. Έχουμε ήδη αναθέσει την έκθεση σε εισηγητή και αυτή η εισηγήτρια δηλαδή θα είναι και η πρώτη ομιλήτρια του σημερινού πρωινού, κυρία Γκαρδίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τον ε, κύριο Επίτροπο για αυτήν την ε, παρουσίαση που μας έκανε για την πρόταση. Σύντομη θα είμαι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Εμείς ε, κατά κάποιο τρόπο έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει νομίζω μεγάλος συντονισμός και σύμπτωση απόψεων μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο κείμενο γίνεται λόγος ε, για συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, τα οποία ε, συζητήσεις οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα οργανώσεις όπως είναι ας πούμε τα ε, νοσοκομεία επιτόπου ε, και τα λοιπά ε, ε, Ήθελα να πω, εκτός από αυτά τα νοσοκομεία υπάρχουν και κάποιες άλλες εξελίξεις σε περίπτωση ας πούμε μεγάλης καταστροφής που ενδεχομένως δεν θα προκύψει ποτέ γιατί είναι, δεν είναι πολύ πιθανή αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί και να συμβεί εάν υπάρχει κάποια πρόβλεψη και για τον, για, την τρομοκρατία. Θα ήθελα γενικώ να καταλάβω πώς η ομάδα εμπειρογνωμόνων διάσωσης ρέσκιου ε, που θα πρέπει να δουν ποια είναι τα επιχειρησιακά μέσα, ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι θα επιτρέψουν την ε, άμεση πρόσβαση στα, μέσα αυτά, πώς, ε, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες, πόσο έχουν προχωρήσει. Αγαπητέ Επίτροπε, καταλαβαίνουμε την αιμονή σας για την πρόληψη και την προετοιμασία και δικιά μας αιμονή και γι' αυτό ε, ε, πραγματικά εκτιμούμε την εργασία η οποία μέχρι τώρα έχει γίνει και την καλή συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν, λέω, να καταλάβω, να κατανοήσω εάν υπάρχουν κάποια επιπλέον input ε, σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε ήδη ε, γιατί η Κομισιόν ε, αναφέρεται εδώ ότι μπορεί να ζητήσει από ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη προετοιμασία συγκεκριμένων μέτρων για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα ήθελα ε, να μου πείτε, αγαπητέ Επίτροπε, εάν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να προβλεφθούν από πλευρά των κρατών μελών κάποιε δαπάνε οι οποίε ενδεχομένω θα χρειαστεί να γίνουν. Και εγώ ως Ιταλίδα γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα κάποια ιστορικά εδάφη, κάποιες ιστορικές περιφέρειες ε, σε συγκεκριμένες ε, καταστροφές και προβλήματα θα πρέπει να προβλέψουμε και την προετοιμασία των κρατών, τα χρήματα τα οποία θα χρειαστεί να καταβάλουν, να δαπανίσουν, ε, τα μέτρα τα οποία θα χρειαστεί να πάρουν, την προετοιμασία την οποία, των υποδομών ενδεχομένως που θα πρέπει να κάνουν. Γιατί καταλαβαίνετε είναι πολλά αυτά που μας απασχολούν και θα ήθελα να καταλάβω λίγο πώς βλέπετε κι εσείς τα θέματα αυτά κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάρλι. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ ε, και που ε, μοιράζεστε μαζί μας αυτές τις λεπτομέρειες. Έχουμε ήδη ε, συναντηθεί, έχουμε συζητήσει ε, και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς ε, συμφωνούμε απολύτως με οποιαδήποτε επιπλέον μέτρα μπορούν να ληφθούν για φυσικές καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη και όλες και τα ακραία φυσικά φαινόμενα τα οποία πλέον είναι πολύ πιο συχνά. Είναι γεγονός και σε αυτό καταλήγουμε όλοι ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο συντονισμένη απάντηση σε αυτές τις φυσικές καταστροφές από όσα είχαμε μέχρι τώρα. Έχω κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν είναι δυνατόν. Η πρόταση αυτή, κατά την άποψή μου, η Rescue, ε, θα πρέπει να ε, αναφέρεται και σε ε, κρατη αλλά και σε ε, χώρες ε, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ακραίο χαρακτήρα, νησιωτικό χαρακτήρα, τις νησιωτικές αυτές χώρες οι οποίες έχουν αν θέλετε διπλό πρόβλημα νησιωτικότητας και απόστασης γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες υποφέρουν από αυτόν τον νησιωτικό χαρακτήρα και και μπορούν πολύ εύκολα να αισθανθούν αποκλεισμένες από οτιδήποτε. Ε, επίσης, και η συνάδελφος αναφέρθηκε σε αυτό, τα νοσοκομεία. η πρόταση είναι αυτά τα field hospitals να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ε, να αναπτυχθούν ε, άμεσα, γρήγορα, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αυτό θα λειτουργήσει. Η Κομισιόν έχει ήδη καταγράψει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο ε, ε, ανάπτυξης γιατί αυτού του είδους τα field hospitals θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσονται εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρλινγκ. Okay. Madame Ευχαριστώ πολύ. Ε, με γούστα και Χαίρομαι, ε, χαίρομαι γιατί μιλάμε εδώ για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ε, που ε, μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα σοβαρά σημαντικά προβλήματα για τους πολίτες της Ευρώπης αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Ξέρουμε ότι η κλιματική αλλαγή είχε ήδη πολλές επιπτώσεις όπως οι πυρκαγιές, το είπαμε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία ακόμα περισσότερο. Επίσης ξηρασία όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία προκαλούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα άμεσα αλλά και έμεσα για όλους τους παραγωγικούς τομείς. Ε, θα ήθελα να ξανασκεφτούμε λίγο πραγματικά τον τρόπο ε, τροποποίησης ε, του πυρήνα του ίδιου του παραγωγικού μοντέλου έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Εγώ θα ήθελα πάντως να υπογραμμίσω κάτι το οποίο ήδη έχει αναφερθεί και το οποίο θεωρώ ότι είναι θεμελιώδους σημασίας. Δηλαδή γνωρίζουμε πλέον, έχουμε επίγνωση της ύπαρξης των κλιματικών προσφύγων που υποχρεώνονται και θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους γιατί πλέον ε, στις ε, χώρες τους, ε, στις περιοχές στις οποίες παραδοσιακά ζουν δεν θα μπορούν πλέον να ζουν. Ε, ήδη από την αρχή του 2018 έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν την Μεσόγειο ε, και αυτού του είδους η ανθρωπιστική κρίση ε, κάνει να τρίζουν τα θεμέλια της ανθρωπιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόσφυγες από την Συρία ήρθαν εδώ γιατί θέλουν να ξεφύγουν από μια εμπόλεμη κατάσταση αλλά να μην λησμονούμε ότι ή πρόκειται και για καταστάσεις οι οποίες έχουν επιδεινωθεί και από την έλλειψη ύδατος. Ε, επομένως κατανοούμε ότι το, το μοντέλο το παραγωγικό το οποίο έχουμε είναι καταστροφικό για τους περισσότερους ανθρώπους. Ήδη ε, το τέλος ε, του 2017 ε, στο περιοδικό Science αναφέρθηκε, υπήρξε ένα άρθρο το οποίο αναφέρει ότι στην ουσία δεν προχωράμε αρκετά γρήγορα, δεν μειώνουμε την επίπτωση των αερίων του θερμοκηπίου και η κατάσταση θα επιδεινωθεί πολύ περισσότερο και μάλιστα αναφέρεται ότι εάν ε, αυξηθεί η θερμοκρασία με πιο γρήγορο ρυθμό τότε μπορεί να αυξηθεί κατά 58% ε, η προσφυγιά λόγω ε, κλιματικών συνθήκων. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και από πολιτική άποψη και επομένω με μεγάλη προσοχή περιμένουμε τα όσα θα λάβει ω μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την έννοια αυτή. Ευχαριστώ. Vielen Dank, Frau Vielen Dank, Herr Kommissar. Äh, für Ihre Ausführungen und für Ihren Vorschlag. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, για την ε, παρουσίαση που μας κάνατε σήμερα αυτής της καλής πρότασης. Ε, όχι μόνο έχουμε προβλήματα λόγω των κλιματικών αλλαγών, αλλά έχουμε και μια ολόκληρη σειρά από άλλες ε, δυσκολίες που επιδεινώνονται περισσότερο λόγω των κλιματικών αλλαγών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω να μου διευκρινίσετε δύο σημεία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο τα εθνικά μέσα να τεθούν στη διάθεση όλων. Σε κάποια συνεδρίαση μου είπαν ότι όταν γίνεται μια καταστροφή στη Ρωσία, ας πούμε, ότι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα. Μα κάτι τέτοιο όμω δεν είναι αποδεκτό. Θα πρέπει να γίνεται ε, πιο γρήγορα αυτή η κατάσταση ε, αυτή η κινητοποίηση ε, γιατί να είναι δύσκολο να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη της Ένωσης ενώ τρίτες χώρες το κάνουν πολύ πιο γρήγορα από μας. Ε, πώς θέλετε επίσης να, να μιλήσουμε για πρόληψη ιδιαίτερα όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ε, κατά πόσο γίνονται οι, αυτές οι πυρκαγιές από δόλο. Δηλαδή όχι μόνο να σβήσουμε τις πυρκαγιές πρέπει αλλά και να τις προλάβουμε. Η Πρόεδρος ευχαριστώ. Gracias, Presidenta. Señor Comisario, Επίτροπε, εγώ θα αρχίσω λέγοντας σας, όπως ήδη είπαμε και στην Ολομέλεια, ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί όχι μόνο θέλουμε να προλάβουμε τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και να τις καταπολεμήσουμε, γιατί ήδη βρίσκονται ε, εδώ, ήδη γίνεται η κλιματική αλλαγή. Ε, το κάθε κράτος μέλος ήδη ε, ξε, αισθάνεται ξεπερασμένο λόγω των χαρακτηριστικών των θεομηνιών που ξεπερνούν τα σύνορα δεν αρκούν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας συνήθως σε σχέση με το μέγεθος των καταστροφών. Γι' αυτό χρειάζεται ένας τέτοιος μηχανισμός. Ε, θέλω να παρέμβω για διάφορα σημεία, αλλά θέλω να επιμείνω Ε, εσείς ε, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι περίοδοι χρονικές. Μιλάμε για ε, πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη, πυρκαγιές στην Νότια Ευρώπη. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα προλάβουμε, να μελετήσουμε τους διάφορους κινδύνους, αλλά και τους πόρους τους συγκεκριμένους για την αντιμετώπιση τους που ήδη υπάρχουν στην κάθε περιφέρεια. Τώρα, μηχανισμός αποζημίωσης θα πρέπει να, ε, να υπάρχει, αλλά πρέπει να το τροποποιήσουμε. Στην πρότασή σας μιλάτε για ε, ταμείο αλληλεγγύη και ήδη σε κάποιε περιστάσει σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στην Ισπανία κυρίως, αλλά και σε άλλες περιφέρειες, οι υπολογισμοί που γίνονται για να δούμε ε, αν και κατά πόσο θα πρέπει να παρέμβει το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι λάθος γιατί υπάρχουν περιφέρειες μεγάλες με μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμού οι οποίες συνήθως πετυχαίνουν τη στήριξη από τις ε, ε, πετυχαίνουν να πάρουν να βοηθηθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης ενώ οι μικρότερες περιοχές οι οποίες όμως είναι πιο αεροκατοικημένες και μπορεί να θεωρούνται και πιο πλούσιες ε, δεν τα καταφέρνουν. Α πούμε, στο, επίσης, στο φυσικό δρυμό της Ρονιάνα στην Ισπανία δεν υπήρξε καμία ε, βοήθεια, ενώ ήταν ένα πάρκο προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποιες αλλαγές αυτόν τον κανονισμό για να κλείσω με μια ερώτηση που αφορά την συντονισμό ανάμεσα στα οικονομικά ε, μέσα αλλά και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κλίμα ε, επηρεάζει την υγεία, ε, την οικονομία, την κίνηση, τη δυνατότητα μετακίνησης. Μήπως θα πρέπει να φτιαχτεί ένα παρατηρητήριο που να συντονίζει όλες τις δράσεις σε θέματα κλιματικής αλλαγής, σε θέματα κλιματικής αλλαγής γιατί νομίζω πως έτσι θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Και έπειτα αυτή η πρωτοβουλία για τα στρατιωτικά ή τα κινητά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία εκστρατείας είναι πολύ καλή ιδέα. Ευχαριστώ. Mr. Peterle. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ευτυχισμένο το νέο έτος, Mr. Commissioner. Preživeli smo težko leto in navajeni smo že na požare, na poplave, na suše, nismo pa imeli še... Κοιτάξτε, ε, ε, ε, πολύ καλή η πρότασή σας, ωστόσο εμείς δεν είχαμε στη Σλοβενία ευτυχώς τέτοιες θεομηνίες. Θα πρέπει ε, όμως η πρόληψη να ε, μεριμνεί για όλες τις πτυχές, ας πούμε, και στην πολοδομία ή στην αρχιτεκτονική, στις μηχανικούς, να ε, υπάρχουν εγγυήσεις για μεγαλύτερη σταθεροποίηση των κτηρίων, γιατί υπάρχουν τέτοια φαινόμενα τόσο έντονα που ε, ε, πολλές φορές ε, δεν τα έχουμε προβλέψει και επίσης πρέπει να προστατεύσουμε το τοπίο, την χωροταξία, τα μνημεία μας. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ποιες είναι οι καινοτομίες που μπορούμε να περιμένουμε σε στα θέματα των δασικών πυρκαγιών που είναι στο καρδιά του προβλήματος. Η δουλειά σας, η δική σας θα πρέπει να δημοσιεύεται και να διαδίδεται πολύ περισσότερο γιατί είναι πολύ θετική και ακριβώς αυτή την Ευρώπη χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Γραμματικάκης. Η πρωτοβουλία σας, ε, κύριε Επίτροπε, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε περιοπτώσεις φυσικών καταστροφών είναι, πρέπει να πω, πολύ αξιόλογη και αξίζει να υποστηριχθεί από όλους μας. Αρκεί το χάσμα που υπάρχει πάντα μεταξύ υλοποίηση και γραφειοκρατίας να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο. Η πρότασή σας, ε, θα μου επιτρέψετε να συνοψίσω, έχει δύο σκέλη από τη μία είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας για την άμεση, το τονίζω άμεση διαχείριση καταστροφών και από την άλλη την επιδίωξη άρτιων στρατηγικών ετοιμότητας και πρόληψης σε όλα τα κράτη. Αυτό το τελευταίο θα μου επιτρέψετε να το υπογραμμίσω, διότι το είπατε κι εσείς, φυσικές καταστροφές θα συνεχίσουν δυστυχώς να συμβαίνουν είναι όμως αναγκαίο να πιεστούν τα κράτη να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευθούν οι καταστροφές που προκαλούνται από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στην πατρίδα μου οι πλημμύρες στη Μάδα της Αττικής. Τέλος θέλω να σταθώ σε μια πτυχή του ζητήματος που είμαι βέβαιος ότι σας έχει απασχολήσει, νησιώτικη καταγωγή είστε κι εσείς όπως κι εγώ και το ανέφερε ήδη με πολύ εύστοχο τρόπο η κυρία Ντάλη. Θεωρώ, κύριε Επίτροπε, ότι είναι απαραίτητο όταν νομοθετούμε μηχανισμούς αλληλεγγύης στην Ευρώπη να έχουμε πάντα στο μυαλό μας την νησιωτικότητα, την ύπαρξη νησιών, μικρών ή μεγάλων. Αλλιώς φοβούμε ότι οι ευεργετικές τους διατάξεις δεν θα φτάσουν ποτέ στους πολίτες των νησιών. Για παράδειγμα, είναι φανερό το κριτήριο του 1,5% του ΑΕΠ για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης είναι προβληματικό για τα νησιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το υπέροχο νησί της Αμοθράκης. Καλό όλους τους συναδέλφους να το επισκεφθούν. Που υπέστη πρόσφατα πρωτοφανείς καταστροφές λόγω πλημμύρας. Το νησί όμως, όπως και πολλά άλλα, έχει την ατυχία να ανήκει σε υπηρετική περιφέρεια, εκείνη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φαντάζομαι το ξέρετε. Είναι συνεπώς αδύνατο να ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο κριτήριο και το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι σποράδες αλλά και άλλα νησιά της Ευρώπης που ανήκουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Το δεύτερο μου παρατήρηση κύριε πίτροπε τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ανταγωνιστικά για τους Δήμους και τις περιφέρειες. Οι νησιωτικοί δήμοι όμως είναι κατά κανόνα πολύ μικροί, με περιορισμένους πόρους και δυσκολεύονται φυσικά να υλοποιήσουν έργα στον τόπο τους. Για την εφαρμογή όμως της πρότασής σας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων. Πώς θα εξασφαλιστεί λοιπόν ότι οι μικροί ευάλωτοι και νησιωτικοί δήμοι δεν θα παραμείνουν αποκλεισμένοι. Τέλος, στο σκέλος της ετοιμότητας και της πρόληψης μια ακόμα παρατήρηση κύριε Επίτροπε. Πώς σκοπεύετε να εμπλέξετε την τοπική αυτοδιοίκηση που καλείται πρώτη να διαχειριστεί τις καταστροφές ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές. Ελπίζω κύριε Επίτροπε και τελειώνω ότι οι αδυναμίες αυτές θα αντιμετωπιστούν και θα μπορούμε όλοι να σας συγχαρούμε για τις προτάσεις και για το μέχρι τώρα έργο σας. Ευχαριστώ. Thank very σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Ορίστε κύριε Επίτροπε, είδατε πόσο ε, έντονο είναι το ενδιαφέρον για το θέμα. Έχετε το λόγο για να μπορέσετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις θετικές παρεμβάσεις και τις ερωτήσεις σας. Να μου επιτρέψετε να απαντήσω ωστόσο στη μητρική μου γλώσσα, έτσι ώστε να μπορέσω να είμαι και ακριβέστερος για τις συγκεκριμένε ερωτήσεις σας. Ξεκινήσω από τις ερωτήσεις της ε, ραμπορτέ της συναδέλφου της κυρίας Γκαρτίνη. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι ένα σημαντικό κομμάτι της πρότασης αναφέρεται και στην αντιμετώπιση των επιδημιών και το ρόλο που θα έχουν τα δικά μας επιχειρησιακά μέσα για νοσοκομεία τα οποία θα είναι mobile hospitals και θα μπορούν να ανταποκριθούν με αμεσότητα σε αυτές τις έκτακτες ανάγκες. Έχουμε ήδη μια εμπειρία, μπορεί κάποιοι από σας να μην το έχετε προσέξει, στα πλαίσια του παρόντος συστήματος υπάρχει το EU Medical Corps. Ήταν αποτέλεσμα και της προσωπικής μου εμπειρίας ως Ebola Coordinator και ήδη έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής αντιμετώπισης προβλημάτων όπως ο κίτρινος πυρετός στην Αγγόλα και απεδείχθη ότι ήταν το καλύτερο lesson learned για μας από την περίπτωση του έπολα. Ε, ώστε υπάρχει μια εμπειρία πάνω στην οποία θα χτίσουμε έτσι ώστε να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί για να στείλουμε αυτά τα κινούμενα νοσοκομεία, τα κινούμενα λάμψ σε στιγμές όπου θα αντιμετωπίζει οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη μας είτε μια φυσική καταστροφή είτε ακόμα και μια επίθεση τρομοκρατική. Ε, υπάρχει σημαντικό εξπερτής, σημαντική γνώση γύρω από αυτό και θεωρώ ότι μαζί με άλλους μηχανισμούς της Ένωσης μέσω ενός συντονισμού θα μπορέσουμε να δράσουμε καλύτερα. Θέλω όμως να διευκρινίσω αυτό που τόνισα εξ αρχής. Rescue is not a replacement. Το rescue δεν αντικαθιστά την πρωταρχική ευθύνη των κρατών μελών. Θα έρθουμε να συμπληρώσουμε αυτή την ευθύνη. Σας έχουμε δώσει ένα ωραίο διάγραμμα, μια πυραμίδα, όπου παρουσιάζει, ξέρω αν το έχετε δει, είναι αυτή η πυραμίδα, πρέπει να το έχετε δει, που παρουσιάζει το rescue, που, ποιο είναι το structure, ποιο είναι, ποια είναι η δομή. Το πρώτο επίπεδο είναι η ευθύνη των κρατών μελών. Το δεύτερο είναι η αναβάθμιση του παρόντος συστήματος, το European Civil Protection Pool, και το τρίτο είναι το rescue, as part of our collective response, όπως έχουμε πει είναι ένα safety net. Ώστε πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό για να αντιληφθείτε ότι οι μηχανισμοί που, θα, που χτίζουμε και θα χτίσουμε και θα βελτιώσουμε δεν θα είναι μαγικές λύσεις αγωνώντας τα εθνικά επιχειρησιακά μέσα. Που σημαίνει θα τα δούμε όλα στη λογική της συμπλήρωσης των εθνικών μέσων. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την θέση ότι prevention and preparedness is the only way. Είναι η μόνη μας ελπίδα να αντιμετωπίσουμε το climate change και θα υπενθυμίσω ότι αυτή η πρόταση δεν είναι απομονωμένη από άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Είμαι σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους μου, Φιλ Χόγκαν και Κορίνα Κρέτσου, που ασχολούνται με τα, structural funds και όπως είπα, το πιο σημαντικό κομμάτι του prevention και του preparedness, ειδικά η χρηματοδότηση, θα προέλθει από τα κονδύλια των διαρθωτικών ταμείων. Ώστε είναι ένας συντονισμός επιτρόπων θα έχω την ευθύνη να συντονίσω τους συναδέλφους μου ακριβώς για να δώσουμε στο κράτος μέλος, στο κάθε κράτος μέλος με βάση τη δική του εθνική, το δικό του εθνικό σχέδιο το πώς θα μπορέσει να αναβαθμίσει την πρόληψη και την ετοιμότητα μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Να πω ένα πράγμα απλό για να γίνει αντιληπτό. Παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα. Συζητείται πάντα ένα θέμα για τις λεγόμενες αντιπυρικές ζώνες εάν είναι έτοιμες κάθε καλοκαίρι πριν από την μάχη κατά των καταστροφών, κατά των ε, πυρκαγιών. Λοιπόν, αυτό θα μπορεί μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και εδώ είναι ο ρόλος που ρώτησε ο κ. Γραμματικάκης να αναβαθμιστεί αυτή η ετοιμότητα σε ό,τι αφορά τις αντιπυρικές ζώνες, οι οποίες είναι εξαιρετικό κομμάτι στην διαχείριση των πυρκαγιών στην κρίσιμη στιγμή. Η κυρία Ντάλη ε, πολύ σωστά ρώτησε και επέμεινε στον νησιώτικο χαρακτήρα και στο πόσο ε, αυτή η πρόταση θα συνδράμει καταστροφές και άλλα προβλήματα στην ε, νησιώτικη περιοχή της, ε, της Υπήρου μας. Ε, όπως γνωρίζετε, εκτός της δικής μου αρμοδιότητας υπάρχουν ε, διάφορα ταμεία που επιχειρούν να καλύψουν αυτές τις μεγάλες ανάγκες στις νησιώτικες περιοχές. Αντιλαμβάνομαι και ξέρω και από την περίπτωση της δικής μου χώρας ότι ναι, δεν είναι επαρκή το ΡΕΣΚΙΟΥ θα, μπορέσει να συμπληρώσει σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών σε νησιώτικες περιοχές κάποια προβλήματα που παραμένουν ανεπίλητα με βάση τις σημερινές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ρωτήσατε κι εσείς για το θέμα των νοσοκομείων. Είπα πριν ότι έχουμε την εμπειρία από το EU Medical Corps. Θα έχουμε μια αναβάθμιση σίγουρα του EU Medical Corps μέσα από το Rescue, γιατί τώρα το πρόβλημα που έχουμε στο EU Medical Corps είναι ότι πάρα, πολλές, πάρα πολλά από τα κράτη-μέλη δεν είναι καν μέλη. Ήταν πάνω σε voluntary basis η συμμετοχή. Ώστε θεωρώ ότι εάν έχουμε το σύνολο των κρατών μελών, όπως επίσης και τα άλλα μέλη που συμμετέχουν στο European Civil Protection Mechanism, όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Τουρκία, Μοντενέκρο, ε, Φύρομ Σερβία θα αυξηθεί η δυνατότητα μέσα από το παρόν σύστημα για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύσκολες απαιτήσει που έχουν οι, οι φυσικές καταστροφές και ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις στην πρώτη φάση που είναι και η πιο σημαντική με την εμφάνιση νοσοκομείων on the ground. Θα συμφωνήσω πλήρως με την κυρία Τόρες για το ότι ναι, ήδη είμαστε μάρτυρες του νέου κύματος προσφύγων εξαιτία της κλιματικής αλλαγής. Το είδα σε όλε μου τι επισκέψει στην Αφρική, στην Ασία, ότι άρχισαν ήδη άνθρωποι και μετακινούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Αιθιοπία που επισκέφθηκα πριν ένα χρόνο. Είναι γι' αυτό που ως Ευρωπαϊκή Ένωση Διαφωνήσαμε και διαφωνούμε ριζικά με την εκτίμηση του, Προέδρου Τραμπ σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή is not a fake news. Είναι γι' αυτό που είμαστε πρωτοπόροι ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Είναι γι' αυτό που θα επιμείνουμε σε όλες μας τις συναντήσεις ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πείσουμε ναι, ότι όλοι μαζί Παγκοσμίω θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, επειδή έχουμε ήδη προχωρήσει πολύ εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμαστε από όλους όσοι πρωτοπόροι, γι' αυτό έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε και από τους άλλους να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση της Συμφωνίας του Παρισιού. Και είμαστε έτοιμοι, και νομίζω υπάρχουν πολλές δηλώσεις πολλών ηγετών των κρατών μελών που πιστεύουν ακόμη και σε ενίσχυση της ίδιας της Συμφωνίας του Παρισιού. Αγαπητέ συνάδελφε, έχουμε συζητήσει και μαζί ακριβώς αυτό το κρίσιμο ερώτημα που θέσατε για τα... γιατί σήμερα τα εθνικά μέσα δεν διατίθενται στις κρίσιμες στιγμές για να αποστείλουν βοήθεια στα κράτη-μέλη. Θα πω το παράδειγμα της Πορτογαλίας που είναι τόσο ε, πριν τρεις μήνες έγινε και όπως είπα και πριν ήταν για μένα ε, πολύ οδυνηρή εμπειρία το τι έγινε εκείνη τη μέρα με την Πορτογαλία, εκείνες τις μέρες. Όταν η Πορτογαλία ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, δυστυχώς υπήρχε red alert σε όλες τις χώρες που μπορούσαν να βοηθήσουν με το να στείλουν Κανατέρ και άλλα μέσα για αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Πορτογαλία τον Οκτώβριο. Εκείνες τις μέρες ήμουν στη Γαλλία, στην Νιμ, ενδεχομένως στο καλύτερο κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών στην Ήπειρό μας. Αλλά όλες, όλα τα reports από όλα τα μήκη και πλάτη της Γαλλίας παραδείγματος χάρη έλεγαν ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει αυτή την σκληρή πραγματικότητα και δεν μπορεί να αποστείλει οτιδήποτε εκτός της Γαλλίας διότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσει για δικές της ανάγκες. Και εκεί, και ως πολιτικοί συζητάμε τώρα, δεν υπήρχε περίπτωση κανείς πολιτικός να αγνοήσει αυτά τα reports από τους ειδικού και να στείλει οτιδήποτε μέσον εκτός της χώρας, είτε από την Ιταλία, είτε από την Ελλάδα, είτε από την Κροατία, είτε από την Ισπανία και αντιληφθήκαμε ότι η Πορτογαλία έμεινε μόνη. Έμεινε μόνη διότι δεν υπήρχε ένας μηχανισμός πάνω από, τις, από τα national capacities και resources, πάνω από τις εθνικές δυνατότητες, έτσι ώστε εκείνη τη στιγμή να μπορέσει να παράσχει τη βοήθεια που δεν μπορούσαν να κρατημέλει. Εκεί ακριβώς είναι ο ρόλος του rescue. Ότι θα ανταποκριθεί τη στιγμή που Όλοι οι εθνικοί πόροι και ικανότητες δεν είναι επαρκείς, ναι. διότι κάθε μια από τις χώρες μέλη μας δυστυχώς και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που είπατε, ότι τα εθνικά μέσα ήταν αδύνατον να σταλούν εκτός από το κάθε κράτος μέλος, διότι δεν μπορούσαν να αγνοήσουν τις δικές τους ανάγκες και εκεί πρέπει να έχουμε αυτό το safety net, το συμπληρωματικό μέσο για να το στείλουμε στην κρίσιμη στιγμή. Γι' αυτό δεν μιλάμε για new γιατί δεν χρειαζόμαστε staff on the ground, το κάθε κράτος μέλος μέσα από τις δικές του εθνικές εθνικούς σχεδιασμούς έχει ικανοποιητικό staff, αλλά αυτό που μιλάμε, παραδείγματος χάρη για, την, ε, για τις πυρκαγιές, είναι ότι θα χρειαστούμε κάποια κανατέρ, κάποια ελικόπτερα, τα οποία θα είναι European Own Capacity, ευρωπαϊκή δυνατότητα για να ανταποκριθεί σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών έχετε δίκιο ότι χρειάζονται πολλά. Και κάπου υπήρξε δόλο. Υπήρχαν περιπτώσει, ναι, που σε κάποιε χώρε για λόγου μη ικανοποιητικού χτιματολογίου, μη ικανοποιητικού ε, συστήματος διαχωρισμού των ε, περιοχών, κάποιοι έβαλαν πυρκαγιέ με στόχο να αυξήσουν τις ε, προσωπικέ του δυνατότητε. Ακριβώ μέσα από το prevention and preparedness τα structural funds θα χρηματοδοτήσουν με τα κράτη-μέλη τέτοιες πολιτικές για να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά και να μην υπάρχει κίνητρο για οποιοδήποτε να προχωρήσει σε τέτοιες δόλιες πράξεις. Για το Solidarity Fund. Το Rescue είναι κάτι ξεχωριστό από το Solidarity Fund. Όπως γνωρίζετε το Solidarity Fund ανήκει στις αρμοδιότητες της συναδέλφου μου της κυρίας Κρέτσου. αυτό που θα πω όμως είναι κάτι απλό και να κάνω μια σύγκριση με το πόσα λεφτά έχουμε εξοδέψει μέσω του Solidarity Fund και ειδικά στις περιπτώσεις των φλάτς, των πλημμυρών στην Κεντρική Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια και αν αυτά τα λεφτά τα χρησιμοποιούσαμε για prevention and preparedness. Είναι σίγουρο από μελέτη ότι θα χρειαζόμαστε λιγότερα λεφτά και θα σώζαμε και ζωές και θα σώζαμε και περιουσίες. Που σημαίνει είναι καλύτερα παρά να δίνουμε λεφτά για το solidarity fund να δίνουμε για το prevention and preparedness. Προς Θεού όμως. <laughs> Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει solidarity fund γιατί αναπόφευκτα δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα που θα χρειαστούν ενίσχυση οι περιοχές. Θεωρώ ότι ε, η συνάδελφος κυρία Κρέτσου πάντα ανταποκρίνεται σε αυτέ τι ειδικέ περιπτώσεις. Έχει ήδη υποσκεφθεί από ό,τι ξέρω και την Γαλήθια και άλλε περιοχέ στην Πορτογαλία για να δει από πρώτο χέρι on the ground και να αξιολογήσει την κατάσταση και να δώσει λεφτά από το Solidarity Fund για αυτές τις περιπτώσεις. Αν υπάρχουν κάτι άλλο μπορούμε να το δούμε σε συνεργασία και να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Αλλά θα επιμένω σε αυτό που είπα. Είναι prevention is better than cure. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Προτιμότερο να δώσουμε τα λεφτά που θα είναι και λιγότερα στο prevention and preparedness παρά να περιμένουμε να τα δώσουμε μέσω του Solidarity Fund. Έχει αποδειχθεί και από μελέτες και στην πράξη ότι είναι η καλύτερη ανταπόκριση εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών. παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής. Ε, είναι, από ό,τι ξέρω από τον συνάδελφο Κανιέτε, υπάρχουν πάρα πολλά ε, υπηρεσίες, στην Ευρω... τα σέρβισες μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούν από πολύ κοντά όλες τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και γι' αυτό, όπως είπα, είμαστε οι πρωτοπόροι μέσω της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Τώρα, εάν θα χρειαστεί να αναβαθμιστεί, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα είναι ανοιχτή σε νέες προτάσεις οι οποίες θα αναβαθμίζουν τη δυνατότητα των υπηρεσιών για να ανταποκριθεί καλύτερα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Έχετε δίκιο, my dear colleague, former Prime Minister, ότι ναι, θα χρειαστούμε να αναβαθμίσουμε την πολεδομία και τη χωροταξία μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ειδικότερα τα structural funds. Και αυτός θα είναι ο ρόλος της συνεργασίας μας με τον συνάδελφο Φιλ Χόγκαν και την συνάδελφο Κορίνα Κρέτσου. Θεωρώ δηλαδή ότι το Rescue θα είναι ακριβώς η ομπρέλα που θα βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά ταμεία να είναι ο βασικός ενισχυτής της πρόληψης και ετοιμότητας μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι through rescue we can demonstrate, θα μπορέσουμε να δείξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Θεσμή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια γραφειοκρατία που όλη μέρα ασχολείται με χαρτιά και έχει ένα πρόσωπο εντελώς μακριά από τις καθημερινές ανάγκες του Ευρωπαίου πολίτη. Έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο και μπορεί να παρέχει χειροπιαστή αλληλεγγύη όταν οπουδήποτε στην Ευρώπη θα έχουμε φυσική καταστροφή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να πείσουμε τις πολίτες μας ότι ναι, η Ευρώπη μπορεί να έχει αλληλεγγύη όταν χρειάζεται ο Ευρωπαίος πολίτης. Ότι δεν είναι όλο αυτό που πιστεύει ο κόσμος ότι είμαστε μακριά από τα καθημερινά του προβλήματα. Και το Rescue είναι το πιο τρανό παράδειγμα χειροπιαστής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα πω το παράδειγμα της δικής μου χώρας όταν αντιμετώπισε πριν δύο χρόνια καλοκαίρι πυρκαγιές οι οποίες ήταν πάρα πολύ καταστροφικές. Μέσω του παρόντος μηχανισμού στάλθηκαν δύο αεροπλάνα, ένα γαλλικό και ένα ιταλικό και αμέσως άλλαξε η διάθεση της κοινή νόμης απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θεώρησε ο απλός άνθρωπος ότι ναι, η Ευρώπη είναι κοντά μας. Μέσω ακριβώς αυτής της βοήθειας εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Και αυτό επιμένω ότι ναι, το rescue θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα προσφέρει βοήθεια σε κρίσιμες στιγμές φυσικών καταστροφών αλλά την ίδια στιγμή αναπόφευκτα, αναφυσβήτητα γίνεται ένα πολιτικό εργαλείο για να στείλουμε το μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες ναι, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν ανθρώπινο πρόσωπο. Σε ό,τι αφορά την Ναι. Ε, για το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων που θέσατε ε, και ήταν ένα θέμα που ζήσαμε αυτή την φοβερή καταστροφή στο Λονδίνο και είδαμε όλοι πόσο σημαντικό θέμα είναι για όλους μας. Ε, γνωρίζω ότι η συνάδελφός μου η Ελίζα Μπέτα δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα και ετοιμάζουν τα σερβίσε μια καινούργια πρόταση που θα έχει σχέση με την ανθεκτικότητα των κτηρίων. Είναι όντω πολύ σημαντικό, αλλά σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του Ρέσκιου σε αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι απλώ μια άμεση ανταπόκριση όταν έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορεί το Ρέσκιου να, υποκαταστήσει άλλα σερβίσε σε νομοθεσίε που αφορούν την ανθεκτικότητα των κτηρίων. Κλείνω ε, με, την ερώτηση του συνάδελφου κ. Γραμματικάκη. Τα σχόλιά σας για το Ταμείο Ελληνικής πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά και για μας. Γνωρίζετε ότι η συνάδελφός μου η κυρία Κρέτσου είναι ενήμερη και πάντοτε διαθέσιμη για συζητήσεις και με τις εθνικές κυβερνήσεις και με τις τοπικές, ε, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες τοπικές ε, ε ε, regional authorities. Ε, υπάρχει μεγάλη συζήτηση πώς θα αυξηθούν αυτά τα κονδύλια. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ενδεχομένω μέσα στο νέο MFF. Είναι συζήτηση που θα γίνει και στα πλαίσια του Κοινοβουλίου και στα πλαίσια του Συμβουλίου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για τον ρόλο των περιφερειών, ειδικότερα στον τομέα της πρόληψης, και σε μερικέ χώρε, όπω τη Γερμανία, αντιλαμβάνεστε ότι η κύρια ευθύνη ανήκει ή στι περιφέρειε. ώστε οι περιφέρειε θα είναι ο βασικό μα σύμμαχο για το prevention και το preparedness. Έχω ήδη ζητήσει να συναντηθώ με την Επιτροπή των Περιφοριών, ενδεχομένω τον επόμενο μήνα, για να ξεκίνησα επαφέ με εκπροσώπου εθνική και τοπική αυτοδιοίκηση σε κράτη-μέλη. Έχω ήδη επισκεφθεί ε, το Ανόβερο, τη Βρέμη και το Αμβούργο ακριβώς για να συζητήσω και σε επίπεδο περιφερειών. Έχω κάνει επαφές με τον ε, Υπουργό στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία χθε και τις επόμενες μέρες θα, ε, σήμερα στη Βουλγαρία με την Βουλγαρική Προεδρία, θα πάω στη Φιλανδία, στη Σουηδία, στη Δανία, όλες τις χώρες περίπου για να μπορέσω ακριβώς να συζητήσω μαζί τους και να βελτιώσουμε ενδεχομένω ακόμα και την πρόταση σε σημεία που αφορούν τι εθνικέ κυβερνήσει και τι τοπικέ αυτοδιοικήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Έχω καταγράψει όλες σας τις ανησυχίες. Πιστεύω ότι σας πρόσφερα κάποιες απαντήσεις έτσι ώστε να πιστείτε ότι το rescue είναι όσο ποτέ αναγκαίο για να αποτρέψουμε μια επόμενη μεγάλη φυσική καταστροφή στην Ευρώπη. Και εκεί όντως θα δείξουμε όλοι μας ότι ναι, η Ευρώπη έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την αποφασιστικότητα που δείχνετε για την πρότασή σας βεβαίως θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας στηρίξουμε και να αντιμετωπιστεί σωστά η κατάσταση με την σωστή προπαρασκευή και προετοιμασία για αντιμετώπιση των θεομηνιών. Ο Επίτροπος, σας ευχαριστώ πολύ και οφείλω να πω βεβαίως ότι είμαι πρόθυμος να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε συνάντηση επιθυμείτε με οποιονδήποτε από εσά αν θέλετε κάποια διευκρίνηση ή βεβαίως να συζητήσουμε και οποιαδήποτε νέα πρόταση που θα μπορούσε να βελτιώσει την πρόταση μου. Πιστεύω ότι η συλλογική σοφία είναι καλύτερη από την ατομική του καθενός. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, λέει η Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα στην αρχή, έχουμε κάνει μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Θα ακολουθήσει τώρα λοιπόν η συζήτηση ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για οι Υπηρεσίες. Δίνω το λόγο στον κύριο Αντρέη Γιάν uh, Good morning, uh, uh, chair. Good morning. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, καλημέρα και στις κυρίες και κυρίους Ευρωβουλευτές σύντομη παρουσίαση. Έχω και μια ε, παρουσίαση με διαφάνειες. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα φάρμακα κυρίως αναφέρεται σε καινοτομία, αλλά χρειάζεται να λυθεί επίσης και η ποιότητα και η ασφάλεια. Οι φαρμακευτικές εταιρείες βέβαια προσανατολίζονται στην αγορά και δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τι ανάγκε των παιδιών. Στόχος λοιπόν του παιδιατρικού κανονισμού ήταν που είναι εφαρμοστείο από το 2007 και πέρσι κλείσαμε τα 10 χρόνια που ε, λειτουργεί αυτός ο κανονισμός. Στην έκθεση που συντάσσουμε και που δημοσιεύσαμε ήδη από τον Οκτώβριο του 2017 έχουμε περιλάβει τα αποτελέσματα των αναλύσεων των επιπτώσεων των πρώτων δέκα ετών της εφαρμογής του κανονισμού και αν θέλετε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια πρόκειται για progress report στην πραγματικότητα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε έναν αριθμό παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή του κανονισμού και να λάβουμε υπόψη και τα όσα ζήτησε στο ψήφισμά του του Σεπτεμβρίου 16 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση δείχνει ότι έχει γίνει πρόοδος, η παιδιατρική έρευνα έχει προχωρήσει, υπάρχουν περισσότερα εγκεκριμένα φάρμακα για παιδιά, με λεπτομέρειες βλέπετε και στην διαφάνεια ότι οι κλινικές έρευνες και δοκιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την έκθεσή μας, άνω των 50 ε, δοκιμών με συμμετοχή παιδιών και είμαστε βέβαιοι ότι θα αυξηθούν κι άλλο όταν θα εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές. Κάνουμε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή <clears throat> ασφάλεια για τα παιδιά με διαφάνεια κλινικές δοκιμές για να ενδυναμωθούν περισσότερο ακόμη τα παιδιά και οι γονείς τους. Στην διάρκεια της περίοδου αυτής είδαμε έγκριση, αδειοδότηση δηλαδή, 260 νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Και οι λεγόμενες PIP ξεπέρασαν τις χίλιες το 2017. Αυξάνεται δηλαδή ο αριθμός τους. Λαμβάνοντας υπόψη ε, την περίοδο αυτή, η περίοδος που είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί η κλινική έρευνα, μπορεί να ε, χρειάζεται και 10 χρόνια και υπάρχει αυξανόμενος αριθμός PIP τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για τα παιδιατρικά φάρμακα με βελτίωση και των φυλαδίων που εγκλείονται στα ε, ε, κουτιά και θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι η μείωση του κινδύνου ε, ε, για τα, από τα παιδιατικά, φάρμακα δεν μπορεί να αφαιθεί μόνο στην νομοθεσία. Επηρεάζεται για από παράγοντες. Για παράδειγμα, επένδυση στις ε, χώρες μέλη. Επίσης, οι παιδίατροι μπορεί να μην αρχίσουν να υιοθετούν αμέσως τα νεοαδιοτηθέντα ε, παιδιατρικά φάρμακα. Η έκθεσή μας μας επιτρέπει να διευκρινίσουμε επίση και σε ποιου τομεί η παιδιατρική έρευνα δεν έχει σημειώσει συγκεκριμένη πρόοδο και ιδίω είδαμε κάποιες βελτιώσεις ότι η ανάπτυξη του παιδιατρικού φαρμάκου εξακολουθεί να ε, βασίζεται στην παράλληλη εξέλιξη φαρμάκων για ενήλικους. Δεν λαμβάνουν δηλαδή υπόψη οι φαρμακευτικές εταιρείε και ιδίως δεν λαμβάνονται υπόψη καρκίνοι σε παιδιά και κάτω των 15 ετών που είναι πολύ σπανιότεροι από ό,τι στους ενήλικους κάτω από το 1% όλων Ωστόσο, είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε παιδιά μεταξύ 1 και 14 ετών. Για το λόγο αυτό, η καρκίνη αυτή, όπως και άλλες αποκλειστικά παιδιατρικές ασθένειες, πρέπει να καλυφθούν από τη σχετική νομοθεσία. Πριν να προτείνουμε οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή στον παιδιατρικό κανονισμό, χρειάζεται να ελέγξουμε καλύτερα ποια είναι η ομάδα συμφερόντων, βιομηχανία, ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, πώς θα συνδυάσουμε τις συνέργειες μεταξύ του παιδιατρικού κανονισμού και των άλλων συναρμόδιων κανονισμών και να διασφαλίσουμε ότι η ισορροπία μεταξύ αυτών με τις διάφορες ρυθμίσεις θα εξακολουθήσει να είναι κατάλληλη για να διευκολύνει την ανάπτυξη και διαθεσιμότητα παιδιατρικών φαρμάκων. Γι' αυτό μέχρι το 2016 είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή τη βελτιωμένη νομοθεσίας, την αξιολόγηση των παιδιατρικών φαρμάκων με νομοθεσία που θα δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν οι κανονισμοί αυτοί. Η έκθεση που έχουμε δημοσιεύσει δεν αρκεί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα περισσότερο, διότι μόνο η συνδυασμένη άποψη των παιδιατρικών ε, των αδερμοδίων για τα παιδιατρικά φάρμακα αλλά και για τα ορφανά φάρμακα για τις ορφανές νόσους δηλαδή θα επιτρέψει την πρόοδο αυτή. Ωστόσο δεν έχουμε λάβει άμεση δράση λόγω έλλειψης ε, σχετικής έρευνας για τους παιδιατρικούς καρκίνους. Η ανάληψη των δράσεων αυτό βλέπετε και στη διαφάνεια μόλις άρχισε για την εφαρμογή του Class Waiver που θα αρχίσει να εφαρμόζεται και πάντοτε σε συζήτηση, σε, διαβούλευση με τους αρμόδιους παιδιάτρους. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν εταιρική ευθύνη που υπερβαίνει το γράμμα του νόμου. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γιατί η συσσωρευμένη γνώση για την ανάπτυξη αντικαρκυνικών φαρμάκων για τους ενηλίκους να μην χρησιμοποιηθεί και εποφελία των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον οργανισμό EMA το 2018 θα οργανώσει εργαστήρια με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να προωθήσει βραχυπρόθεμες δράσεις για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα παιδιατρικών φαρμάκων. Η εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών, το τονίζω αυτό, είναι κρίσιμη. Το προωθούμε αυτό και σε διεθνές επίπεδο με στενές επαφές με το FDA των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στο Λονδίνο μάλιστα διεξήχθη ειδικό εργαστήριο για να συνεργαστούμε μαζί με τους εκπροσώπους του FDA και να προωθήσουμε από κοινού την ατζέντα αυτή. Ολοκληρώνοντας, ας μην λησμονήσουμε δύο άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν το δυναμικό να ενισχύσουν την έρευνα στο παιδιατικό φάρμακο. Πρώτον για τις σπάνιες ασθένειες, εκεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για περίπλοκες και σπάνιες νόσους που αποτελεί και πλατφόρμα για την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών και για την ε, knowledge sharing και τη διευκόλυνση της χρήσης μεγάλων όγκων δεδομένων μπορεί σε αυτά να βασιστεί και η προσπάθεια πρόθεσης νέων ιδεών για ασθένειες που εκτυπούν τον παιδικό πληθυσμό και για καρκίνους και εκεί συνεργαζόμαστε στενά με τον οργανισμό EMA. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τα λόγια μου και αναμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Να δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους που το ζήτησαν. Η κυρία Γκροστέτ πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι πολύ ικανοποιημένοι που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μετά από την παρουσίαση της έκθεσης της Επιτροπής ε, ε, και περίμενα την έκθεση αυτή εδώ και καιρό. Πιστεύω πως χάσαμε πολύ χρόνο και είμαι ευτυχής που υπάρχουν διάφορες προτάσεις και να θυμίσω ότι ο κανονισμός, μάλλον και διαπιστώνουμε ότι εν μέρη ε, πέτυχε τους στόχους του αυτός ο κανονισμός, όχι όσο θα το θέλαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει η έκθεση της Επιτροπής ε, θεωρώ πως ε, κάνει μια σωστή διάγνωση της κατάστασης. Λυπούμε μόνο που η, ε, δεν είναι πιο συγκεκριμένες οι λύσεις που προτείνει. Αν και γίνονται κάποιες προτάσεις. Κάποια στοιχεία λοιπόν περιλαμβάνονται στο κοινοβουλευτικό ψήφισμα που ψηφίσαμε πέρυσι, όπως η έλλειψη της εξέτασης του μηχανισμού για τα διάφορα ε, ε, μόρια. Όταν δηλαδή τα εργαστήρια αποφασίζουν ή όχι να προχωρήσουν σε εμπορευματοποίηση ε, μιας εφεύρεσής τους. Επίσης για τον παιδικό καρκίνο είναι ένας θεραπευτικός τομέας που έχει πολύ αφαιθεί στην άκρη και υπογραμμίζει αυτό τα ελλείψεις της εφαρμογής του κανονισμού, δηλαδή παιδιατρική ανάπτυξη, καθαρά παιδιατρική, δηλαδή που να μην συνδέεται με πρόγραμμα για τους ενήλικες. Συχνά όταν η ε, ε, ασθένεια δεν έχει, δεν έχει χτυπήσει ενήλικες δεν υπάρχει θεραπεία για τα παιδιά. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει περισσότερο να, να πολεμήσουμε για την χρήση των ε, φαρμάκων αλλά και ε, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχουν δημιουργηθεί σαφές, σαφείς παροτρύνσεις και κίνητρα αλλά θα πρέπει να είναι πολύ πιο καλά σταθμισμένες για να ευνοηθεί ακόμη περισσότερο η παιδιατρική αγωγή. Ε, η Κομισιόν πρέπει να εμβαθύνει περισσότερο στον κανονισμό για τα παιδιατρικά φάρμακα αλλά και τον κανονισμό για τα φάρμακα τα ορφανά σε συνδυασμό δηλαδή Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει ακόμα να αναπτυχθούν. Θα εφαρμοστεί, θα γίνουν και ατελειέ, δηλαδή ε, σεμινάρια, θα υπάρξει δηλαδή συνεργασία ανάμεσα στους παιδιάτρους της την Κομισιόν και ελπίζω και το Κοινοβούλιο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε ε, μένω ε, σε επιφυλακή ώστε να μπορέσουμε όσο γίνεται με καλύτερο τρόπο να ε, ολοκληρώσουμε αυτή την εξέταση και να ε, καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Η κυρία Καμπεθόν, ευχαριστώ. Θέλω να, να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την τοποθέτησή της, για την επικοδομητική αυτοκριτική που άσκησε ε, και για την έκθεση που μας υπέβαλε. Βεβαίως αυτός ο κανονισμός δίνει περισσότερες άδειε για τα φάρμακα, αλλά όχι για τα παιδιά. Για τα παιδιά είναι σπάνιο. Όπως λέει και η έκθεση της Κομισιόν, τα νέα φάρμακα για τα παιδιατρικά φάρμακα ορίζονται από τις ανάγκες των ενηλίκων. Έχουμε λιγότερο προχωρήσει όσον αφορά την προτεραιότητα και την ανάγκη τη συγκεκριμένη που έχουν τα παιδιά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, δούμε πώς γίνεται η τοποθέτηση. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να περιοριστεί το θέμα της διάθεσης ε, παιδιατρικών φαρμάκων, να δούμε ε, εφόσον υπάρχουν μηχανισμοί για έρευνα. Και Εν πάση περιπτώσει να εστιάσουμε περισσότερο την έρευνα στις προτεραιότητες που είναι σημαντικές για τα παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι το σημερινό πρότυπο για τα κίνητρα δεν έχει ε, μεγάλη διαφορά από το προτινόμενο. Πρέπει να δώσουμε νέα πρότυπα για έρευνα όταν έχουμε να κάνουμε ε, ε, με τόσο περίπλοκες αρρώστιες όπως ο παιδικός καρκίνος να δώσουμε περισσότερα χρήματα για την έρευνα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει περισσότερες δυνατότητες να θεσπίσει τις δικές της προτεραιότητες. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια σαφή προτεραιότητα που είναι ο παιδικός καρκίνος. Από αυτή την έκθεση επίσης προκύπτει ότι ο κανονισμός για τα ορφανά φάρμακα, δεν ξέρουμε γιατί, δεν είναι αποτελεσματικός για να αναπτυχθούν περισσότερα φάρμακα για τα παιδιά. Ίσως γιατί η αγορά ε, για τους ενήλικους είναι μεγαλύτερη από αυτήν των παιδιών. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί ο σχετικό κανονισμό γιατί πιστεύω πως θα πρέπει να περιοριστεί κάπως ε, η αποκλειστική ε, έρευνα για τους ενήλικες, γιατί πιστεύω πως έτσι θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα αυτός ο κανονισμός για τα παιδιά. Νομίζω πως θα πρέπει να αναθέσουμε αυτή την ευθύνη στην βιομηχανία και ίσως να γίνουν και περισσότερες έρευνες για, ε, ειδικά για τα παιδιά, να υποχρεωθούν δηλαδή οι ε, να κάνουν συγκεκριμένες μελέτες και συγκεκριμένες έρευνες για τα ίδια τα παιδιά. Τέλος, ε, για την εμπορία παιδιατρικών φαρμάκων, νομίζω πως μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει καρπού σε αυτό, αλλά πρέπει να διερευνήσουμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα γιατί θα ήταν ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και το νούμερο των αδειών. Ευχαριστώ. Λίζε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση και για την υποβολή βεβαίω του εγγράφου της εκθέσεως. Πολλοί βέβαια συζητούν τι θα πρέπει να ρυθμίζει η Ευρώπη και τι όχι. Για τα ε, παιδιατρικά φάρμακα είτε θα υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία είτε δεν θα υπάρξει απολύτως καμία πρόοδος. Είναι περιορισμένη η αγορά αυτή και γι' αυτό είναι αναγκαίο να γίνει ευρωπαϊκή συνεργασία και στην έρευνα και στην πρόθεση των ε, ε, παιδιατρικών φαρμάκων και στις συγκεκριμένες θεραπείες. Αυτό οφείλει να το τονίζει κανείς διαρκώς. Και θα πρέπει να είναι σαφές και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέραν αυτής. Θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ την Φρανσουάς Γκροστέτ που υπήρξε η εισηγήτρια για θέματα παιδιατρικών φαρμάκων και, όντοτε, και όντως έχουν γίνει πολλά πράγματα από τότε. Υπάρχουν πολλά παιδιατρικά φάρμακα τώρα που χωρί τον συγκεκριμένο κανονισμό του 2007 δεν θα είχαν υπάρξει. Αυτό είναι η καλή πλευρά τη ιστορία αυτή και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και να το καταστήσουμε σαφέ και προ τα έξω. Θα είναι σωστό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει και ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα. Α πούμε, οι αριθμοί είναι μεν ενδιαφέροντε, αλλά πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, τα ε, παιδιών τα οποία θεραπεύτηκαν ενώ πριν από 10 χρόνια χωρίς τον κανονισμό δεν θα είχαν την ευκαιρία να θεραπευτούν. Τώρα υπάρχει και η μεγάλη βέβαια αρνητική πλευρά, ιδίω για θέματα παιδικών καρκίνων, όπου έχει γίνει πολύ μικρή πρόοδος. Εδώ νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει οποιαδήποτε έκκληση προς την βιομηχανία. Στη βιομηχανία ίσως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με καλή θέληση που να θέλουν κάπως να βοηθήσουν, αλλά εν τέλει οι μέτοχοι των εταιριών αυτών θέλουν να δουν κέρδος και χωρίς κέρδος δεν θα γίνει τίποτα και στον χώρο του παιδιατρικού φαρμάκου. Ας μην είμαστε αφελείς λοιπόν η βιομηχανία έχει ως σκοπό το κέρδος. Είτε λοιπόν οι συνθήκες πλαίσια θα είναι τέτοιες που θα επιτρέπουν αποκομιδή κέρδους από το παιδιατικό φάρμακο, είτε δεν θα γίνει τίποτα. Γι' αυτό και πρέπει να επιβάλλουμε κάποια πράγματα. Ε, είμαι κάπως επιφυλακτικός ε, σχετικά με το εάν πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Ίσως μπορεί να γίνει με συστάσεις του EMA. Όμως, τις προδιαγραφές για τις συστάσεις, συστάσεις αυτές θα πρέπει να τις κάνουμε εμείς, ώστε αυτοί που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην κατεύθυνση αυτή τη φαρμακοβιομηχανία να μπορούν να πείσουν και τους μετόχους τους. Τέλος, γνωρίζω ότι η Γενική Διεύθυνση Σαντέ δεν είναι η αρμόδια, αλλά η Κομισιόν είναι ένα ενίο σύνολο και γι' αυτό θα πρέπει να προωθηθεί και η έρευνα. Υπάρχουν κάποια πράγματα, δηλαδή να τονωθεί ο ρόλος αυτών που ασχολούνται με την έρευνα, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσει. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να βοηθήσουν καλύτερα τα παιδιά που δεν έχουν σχέση με νέα φάρμακα οι δυνατότητες αυτές, αλλά για παράδειγμα με την χρήση υφιστάμενων φαρμάκων, με λιγότερη χημειοθεραπεία για παράδειγμα, για να έχουν τα ίδια αποτελέσματα με λιγότερη χημειοθεραπεία σε παιδιά. Για αυτό το λόγο όμως, για να γίνουν τα πράγματα αυτά, χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Οι χώρε από μόνε του δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την έρευνα αυτή. Πρέπει να δοθεί χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να αναλάβουν οι ίδιε χώρε μέλη και όμω τα χρηματοδοτούμε και εμεί. Αλλά σε ό,τι αφορά την υγεία των παιδιών, εκεί χρειάζεται ανάληψη ευρωπαϊκή δράση. Και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει προτεραιότητα τη ευρωπαϊκή έρευνα και ή δυνατόν άμεσα. Και πάντως το αργότερο όταν θα εγκριθεί το νέο ερευνητικό πρόγραμμα. Αν δεν καταφέρουμε εμείς να ενισχύσουμε την έρευνα για, την, για τον παιδιατρικό καρκίνο, δεν θα μπορέσουν να τα αποκριθούν οι χώρες μέλη. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη. Οφείλουμε να επιταχύνουμε ώστε να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στην έρευνα για τον παιδιατρικό καρκίνο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Κομισιόν που παρουσίασε την έκθεση αυτή σχετικά με την πρόοδο που έχει γίνει για τα παιδιατρικά φάρμακα τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι θετικό το γεγονός ότι ακούμε ότι έχει γίνει πρόοδος όσον αφορά το θέμα αυτό. Ακούσαμε για τις αδειοδοτήσεις που έχουν δοθεί σε νέα παιδιατρικά ε, φάρμακα ε, Λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για έναν κανονισμό που πραγματικά βοηθάει τα παιδιά ε, ε, να έχουν πρόσβαση σε κάποια είδη ε, φαρμάκων. Ωστόσο, όταν αναφερθούμε σε σπάνιες ασθένειες τότε, και τον καρκίνο, τότε τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να βρουν λύση. Επίσης ε, πρέπει να αναφέρουμε ε, ότι υπάρχουν πολλές ε, πρόοδοι όσον αφορά τις θεραπευτικές διαδικασίες για τις παιδικές ασθένειες, αλλά ιδιαίτερως θα πρέπει να σκέψουμε πάνω στις ασθένειες, τις σπάνιες ασθένειες των παιδιών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε όσον αφορά ιδιαιτέρως τα παιδιατρικά φάρμακα για τις ε, ε, σπάνιες ασθένειες. Ε, χρειάζεται μεγαλύτερη, περισσότερη έρευνα, οπωσδήποτε, όμως χρειάζεται ταυτόχρονα και μεγαλύτερος συντονισμός ανάμεσα στους ερευνητές, της, την, την, βιομηχανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η πρόσβαση στην θεραπεία, θεραπευτικές διαδικασίες για τον καρκίνο καρκίνο και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε γιατί αυτού του είδους ε, οι θεραπείες ε, για ε, καρκίνους παιδιών δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ όσο για τους καρκίνους των ενηλίκων. Τουλάχιστον όχι τα τελευταία δέκα χρόνια θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν την άποψή της για το θέμα αυτό. Πρόσφατα ακούσαμε ότι οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των καρκίνων των παιδιών, αλλά οι ερευνητές αυτοί ε, σκοντάφτουν πάνω σε πολλά προβλήματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ε, και τα προσκόμματα όσον αφορά τα παιδιατρικά φάρμακα. Ε, αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και επομένως, όπως είπαν και προηγούμενοι συνάδελφοι, νιώθω πως η Κομισιόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την επιρροή της ε, αλλά και τον χρόνο ε, που έχει ε, μείνει ακόμα διαθέσιμος έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των παιδιών σε παιδιατρικά αντικαρκυνικά φάρμακα αφενός αλλά και γενικότερα ώστε να αναπτυχθεί μια κατάσταση όπου κυρίως για τις σπάνιες ασθένειες να υπάρξει η κατάλληλη έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Κομισιόν ε, για την εισήγηση αλλά και για την αυτοκριτική που έκανε ε, γιατί καταδεικνύεται νομίζω και από τα λεγόμενά της ε, η ανάγκη περισσότερων επενδύσεων στην έρευνα έτσι ώστε να βρεθούν φάρμακα για τα παιδιά. Από αυτή την άποψη μπορώ να ε, συμφωνήσω απολύτως με αυτό που είπε ο συνάδελφος Λίζε, δηλαδή ότι αυτή θα πρέπει να ε, ε, γίνει πραγματική προτεραιότητα της δραστηριότητάς μας. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα τα οποία είπαν ήδη άλλοι συνάδελφοι. Όμως πραγματικά θέλω να υπογραμμίσω ένα στοιχείο και να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ε, προκύπτει ε, διάσταση μεταξύ των παιδιατρικών φαρμάκων γενικότερα και των φαρμάκων για τις σπάνιες ασθένειες αφετέρου. Πολύ συχνά τα φαρμακευτικά εργαστήρια ε, δεν ασχολούνται με τα ε, φάρμακα ε, για τις σπάνιες ή λεγόμενες ορφανές ασθένειες Επίσης, ε, το ε, ε, σχέδιο το οποίο καλύπτει την συνολική οικογένεια των CPC, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες θεραπευτικές υποχρεώσεις, ενώ, για τις περιπτώσεις των σπανίων ασθενειών έχουμε μονάχα την προστασία ως φάρμακο και όχι ως οικογένεια φαρμάκων. Θα πρέπει να αλλάξει η κινητροδότηση όσον αφορά τα παιδιατρικά φάρμακα για τις σπάνιες σπάνιες ε, ασθένειες. Τι κάνει η Κομισιόν για το θέμα αυτό, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αν θέλει να ξαναπάρει το λόγο, παρακαλώ κύριε Ρίση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, που έλαβε χώρα. Όπως είπε και η κυρία ε, Γκροστέτ, το εργαστήριο είναι ανοιχτό και για τους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες θα, τις, θα σας τις δώσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό που ακούστηκε προηγουμένως για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε το μοντέλο της έρευνας. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε λοιπόν ότι εμείς ε, ήδη μέσω του ορίζοντα 2020 χρηματοδοτούμε τέτοιου είδους ε, προγράμματα ε, και πρωτοβουλίες για καινοτόμα φάρμακα. Έχουμε επίσης ένα αρκετά ισχυρό παιδιατρικό ε, δίκτυο το οποίο προσπαθεί να φέρει σε επαφή ε, αυτούς που ασχολούνται με τις ε, κλινικές δοκιμές έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία συνδέονται με την έρευνα. Ο Δ. Λίζε ρώτησε εάν μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα, ε, δηλαδή τι αλλάζει όσον αφορά την πρόσβαση στις, ε, στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν κατάλογο λοιπόν με τα καλύτερα παραδείγματα όπου θα αναφέρονται οι βέλτιστες πρακτικές και οι μελέτες και οι στάντες τις οποίες έχουμε βασιστεί. Σωστά ρωτάτε εάν ε, υπάρχουν αρκετές ε, ε, πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν την βιομηχανία να συμπορευτεί μαζί μας σε αυτήν την διαδικασία. Κοιτάξτε, υπάρχουν νέα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκου, τα Primes, έτσι ώστε ε, να ε, έχουν και οι βιομηχανίες κίνητρο ε, για να προχωρήσουν στην έρευνα έτσι ώστε να προκύψουν νέα φάρμακα και μάλιστα με γοργότερο ρυθμό. Όσον αφορά την έρευνα για τις σπάνιες ασθένειες, πριν από μερικές εβδομάδες η Κομισιόν ε, δημοσίευσε μια νέα πρόσκληση εξειδικευμένη ε, για τις σπάνιες ασθένειες ε, διαδικασία που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευελπιστούμε ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα να προκύπτουν από αυτήν την πρόσκληση και ότι τελικά το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει καλά. Όσον αφορά αυτό που είπε η κυρία Νταλή για τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή η έρευνα μπορεί να προωθήσει τον κανονισμό, μα αυτό είναι ουσιώδες ε, σημείο. Πώς ε, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η διαθέσιμη έρευνα ε, μέσω δημιουργίας δικτύων, μέσω βελτίωσης των υποδομών και να έχει θετική επίπτωση ένα από τα κεντρικά ερωτήματα τα οποία θέλουμε να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση είναι ακριβώς αυτό το θέμα ε, του συνδυασμού των δύο κανονισμών ε, και ε, να δούμε το κατά πόσο, να αξιολογήσουμε το κατά πόσο ο συνδυασμό των δύο κειμένων, των ε, δύο κανονισμών μπορεί να βοηθήσει ή όχι και εάν μπορεί πραγματικά να αυξηθεί, να βελτιωθεί η πρόσβαση ασθενών ειδικών αναγκών σε φάρμακα. Το 19 προβλέπουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να επανακάμψουμε με πολύ συγκεκριμένες ε, προτάσεις και πολύ συγκεκριμένα ε, στοιχεία όσον αφορά τους κανονισμούς αυτούς. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τα όσα υπόθηκαν εδώ. Τώρα πρέπει να ανασκουμποθούμε. Είναι ώρα για δουλειά, είναι ώρα για δράση έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα ε, και να δουλέψουμε ε, για το καλό των ε, ασθενών. Αλλά για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που σας συνόδευσαν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Τώρα έχουμε ένα άλλο σημείο στη σε διάταξη. Μηχανισμοί ελέγχου των ε, εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πλευρά των κρατών μελών. Και δίνω το λόγο αμέσως ε, στον συνάδελφο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει τώρα να ε, λάβουμε θέση σε μια πρόταση της Επιτροπής ε, που τροποποιεί τους κανόνες που και τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τους ελέγχους από πλευράς ε, των κρατών μελών των, των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, Ένω, της Κομισιόν. Δηλαδή, αυτό στόχο έχει να, να, να, να καλύψει κάποια έλλειψη απάντηση από πλευράς ε, των κρατών μελών για κρίσιμα κάποιες φορές θέματα. Να θυμίσω τα όσα είπε ο Πρόεδρος Ζαν Κλοντ Γιούνκερ τον Σεπτέμβριο του 2016. Όλοι ακούσαμε και ε, ε, είμαι βεβαία ότι συμφωνούμε με τα όσα είπε ο Επίτροπος με στόχο να καταγγείλει τη στάση των κρατών μελών που σε πολλές περιπτώσεις δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και επιβάλλουν στη Κομισιόν να το κάνει στη θέση τους. Δυστυχώς από τότε που φτιάχτηκε αυτή η ε, θέση έχουμε, έχει, έχει εμπλακεί το ζήτημα και αυτή η κρίση οδηγεί, δείχνει μάλλον πόσο αδύναμο είναι το σύστημα και ε, περιπλάκει και η συζήτηση η οποία στην αρχή θα ήταν υποτίθεται μόνο τεχνικής φύσης και αυτό θα πρέπει να το ε, έχουμε στο νου μας για το μέλλον και οι προτάσεις της Κομισιόν πιστεύω ότι προχωρούν στη σωστή κατεύθυνση και επιτρέπουν καλύτερη, ε, περισσότερη ευθύνη και υπευθυνότητα για τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, κάποιο στοιχείες μπορούν ακόμα να βελτιωθούν, κυρίως όσον αφορά τη διαφάνεια. Αυτό που θα ήθελα εντόνως να προωθήσω σε αυτήν την έκθεση. Είμαι μάλιστα πεπισμένη ότι για σημαντικά θέματα όπως η φορολόγηση, η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια ε, της, ε, των τροφίμων και η προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο μπορούν αλλά οφείλουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στα κατημέλη και να τα γνωστοποιήσουν και στους, ε, στους πολίτες. Και μόνο ενισχύοντας αυτή τη διαφάνεια και ενημερώνοντας καλύτερα για την διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό το λόγο προτείνω μία διάδοση των ψηφοφοριών τόσο για των επιτροπών όσο και ε, των επιτροπών ε, ε, των αρμόδιων με επεξήγηση ψήφου των κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης να γίνει εξαρτίας ενημέρωσης ευρύτερε για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την ανάλυση των ε, κινδύνων καθώς και την κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα επίσημα ε, επιστημονικά όργανα ε, της Ένωσης, της, τους οργανισμούς της Ένωσης και τους θεσμούς της Ένωσης καθώς και τα κατημέλη. Το ότι θα Δημοσιεύονται οι ψηφοφορίε και τα κράτη-μέλη θα μπορούν να κάνουν και επεξηγήσει ψήφου. Επιτρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, ότι δηλαδή ακόμα και αυτοί που, κάνουν, που απέχουν να μπορούν να εξηγήσουν τη στάση του. Υπάρχει μεγάλη διαφορά αν κανείς λείπει ή αν κανείς απέχει. Ε, είναι μια πολιτική επιλογή αυτή, αλλά δεν θα πρέπει παρόλα αυτά να παραλύει το σύστημα, πράγμα που συμβαίνει αρκετά συχνά τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό και στηρίζω την πρόταση της, της Κομισιόν στο θέμα αυτό. Όμως προσοχή, πρέπει να είμαστε φρόνιμοι στις προτάσεις μας και συνετοί, ώστε να μην αποσταθεροποιηθεί τελείως ένα σύστημα που θυμίζω στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων λειτουργεί. Ε, τέλος, ε, για να σεβαστούμε τη δημοκρατία θα πρέπει να εξασφαλίζουμε την ε, ταυτόχρονη ενημέρωση του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο και αυτό σε όλες τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στους Κιώδης. Η κυρία ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις εξηγήσεις της συναδέλφου και είναι σημαντικό να το συζητήσουμε. Και σε σχέση με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και με, το, με τη γλυφοσάτη έχουμε ήδη κατ' επανάληψη ζήσει τέτοια μπλοκαρίσματα στο παρελθόν. Τα πιο σημαντικά λέχθηκαν ήδη. Αφενός χρειάζεται διαφάνεια στη διάρκεια ολόκληρης διαδικασίας, γιατί το βλέπουμε ξανά και ξανά στις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων να εκφράζονται άλλες απόψεις από αυτές που ακούγονται στις χώρες. Βλέπουμε και πολλές πολιτικές τακτικές κινήσεις εδώ που δεν επιτρέπουν εν τέλει να αντιληφθούμε ποια είναι η πραγματική θέση των χωρών μελών. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή της κατάστασης έτσι. Διότι οι αξιωματούχοι ακολουθούν τις εντολές τους και μετά έρχονται οι υπουργοί και τα τονίζουν ξανά στα Συμβούλια Υπουργών. Εγώ νομίζω ότι σε ολόκληρη τη διαδικασία πρέπει να εμπλακεί η κοινή γνώμη, δηλαδή πρέπει να μπορεί να, να παρακολουθεί. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προδοθεί το, το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών με αιτιολογημένη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου για κατάθεση τροπολογιών. Θα υποβάλουμε τις ορισμένες, αλλά πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Διότι ναι μεν λειτουργήσε το θέμα έως τώρα, αλλά όπου υπάρχουν προβλήματα η λύση τους έχει αναβληθεί. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κινητοποιηθεί αν δεν θέλει να την βαρύνει τελικά η ευθύνη. Κύριε Γκέρλινγκ, ευχαριστώ την εισηγήτρια πρώτα για την εργασία της, διότι τα λέει τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Και συμφωνούμε και εγώ και η πολιτική μου ομάδα υπάρχει μια αμφισημία την οποία διατύπωσε και η ίδια για αυτή την δευτεροβάθμια επιτροπή και είναι σωστό να υπάρξει κάποια ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής αυτής γιατί στις χώρες μέλη να μπορούν να αλλάξουν τη θέση τους μετά. Δηλαδή μπαίνει ένα ακόμη επίπεδο συζήτησης για να μπορέσει να διαμορφωθεί ευκολότερα μια συνένεση. Πάντως το ερώτημα θα είναι, εάν η αλλαγή στην μέθοδο ψηφοφορίας που είναι και το βασικό, αν αυτό αποδώσει, τότε δεν είναι και αναγκαία η δευτεροβάθμια επιτροπή. Είναι λιγάκι δηλαδή σαν να στοιχηματίζει κανείς σε δύο άλογα στον ίδιο αγώνα. Πάντως θα συζητηθεί μεταξύ των σκιωδών εισηγητών το θέμα για να δούμε τι θα προτείνουμε ακριβώς. συμφωνώ ότι δεν πρέπει να καταργήσουμε το σύστημα ούτω ή άλλω πρόκειται το 2% και η επιτροπολογία δεν αποδίδει πάντοτε, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσω και με την τελευταία παρατήρηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της, ε, ε, συγγνώμη, τη συγχύτρια. Και για τον τρόπο αλλαγή τη ψηφοφορία που εγώ νομίζω ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Και πάντω το ελπίζω. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θυμάμαι τα όσα ακούσαμε από τον πρόεδρο ε, Γιούνκερ που εκνευρίστηκε, ε, το λιγότερο που μπορώ να πω, με τα κράτη-μέλη ε, που, που κρύβονται, που δεν ε, θέλουν να πάρουν αποφάσεις ε, και που τελικά ρίχνουν πάντα το μπαλάκι στην Κομισιόν. Αυτά γίνανε στην ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι πολύ σωστά αντιμετωπίζει το θέμα η κυρία Ντελαέ. Ίσως μπορούμε να προτείνουμε δε ακόμα πιο ορθολογικές και λογικές λύσεις γιατί και για θέματα ας πούμε ε, ασφάλειας τροφίμων με εμβληματικότερο θέμα το θέμα της γλυφοσάτης ε, ε, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη κρύβονται τελικά επομένως συμφωνώ απολύτως με την μέθοδο υπολογισμού οπωσδήποτε η μέθοδος υπολογισμού είναι ο ακρογωνιαίος λήθος αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν και πολιτικοί τρόποι επίλυσης Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα απόφασης θα πρέπει οι κυβερνώντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η ευελιξία ε, της εισηγητρίας ε, σε πολιτικό, ε, στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και είναι και πολύ καλή τρίπλα κατά κάποιο τρόπο που έκανε η εισηγήτρια και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα αυτό και βεβαίως η διαφάνεια και βεβαίως η επικοινωνία γιατί τελικά εμείς ε, ε, συνέχεια πρέπει να υπενθυμίζουμε τα πιο αυτονόητα από τα αυτονόητα. Ε, φυσικά διαφάνεια, γιατί φυσικά οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τα θέματα των οποίων υπεραμείνονται οι οι επικεφαλής τους όσον αφορά την ιδέα ε, να πιέσουμε ε, το Συμβούλιο να ληφθεί απόφαση, τι να σας πω, εάν ε, οι εκπρόσωποι δεν έχουν βρει την δυνατότητα συμφωνίας, συνένεσης στη διάρκεια της, και στη διαδικασία της ψηφοφορίας, δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να πιέσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ μπορώ να συμφωνήσω με το σύνολο των προτάσεων. Σας ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. Η κυρία Χόκη από την ε, Κομισιόν. Ή κάποιος άλλος, όποιος θέλει. Η, η κυρία Ντελαέ πήρε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων που πήραν το λόγο. Μόνο οι γυναίκες πήραν το λόγο. Ε, ίσως αυτό είναι και ένα σημάδι Ε, πρόεδρος, θα ήθελα πρώτα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν και μετά θα σας δώσω το λόγο. Ω, συγγνώμη, λέει κύριε Δελαέ. συγγνώμη. Η Κομισιόν παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Άκουσα ε, γενικά πολύ ε, ε, στήριξη και από την εισηγήτρια πρωτίστως αλλά και από τους υπόλοιπους βουλευτές όσον αφορά το πνεύμα και τον προσανατολισμό της πρότασης της Κομισιόν η οποία θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα οποτεδήποτε ένα πρόβλημα παρουσιάζεται. Δεν θέλουμε ε, να αμφισβητήσουμε συνολικά το σύστημα. Καθόλου δεν είναι ο στόχος μας ή η πρόθεσή μας αυτή. Διαπιστώνουμε επίσης ε, και ε, υποστήριξη για τις τροπολογίες οι οποίες αφορούν την διαφάνεια δράτω με δε της ευκαιρίας. Για να εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί μία από τις τροπολογίες αφορούσε την ταυτόχρονη πληροφόρηση Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ήδη ε, αυτό διασφαλίζεται από τον κανονισμό ΚΑΝΤ και επομένως ε, ταυτόχρονα τα στοιχεία φτάνουν και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πλέον διασφαλισμένο. Προέκυψε μια ερώτηση γιατί χρειαζόμαστε το Συμβούλιο όταν ε, η όταν λειτουργούν οι διάφοροι ε, τρόποι πλειοψηφικής ε, ψήφου. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα may στα αγγλικά, στη διατύπωση, ε, επομένως είναι προαιρετικό και μπορεί να προχωρήσουμε σε δεύτερο γύρο επιτροπολογίας, διαδικασίας επιτροπής δηλαδή. Και ερώτηση γιατί το Συμβούλιο πρέπει να παίξει ρόλο εδώ. Απάντηση, μα γιατί ακριβώς εκεί βρίσκονται ε, όλα τα κράτη-μέλη γύρω από ένα τραπέζι ε, σε ε, θέματα τα οποία, για τα οποία η Κομισιόν ελέγχεται από τα κράτη-μέλη, ούτε όχι καν από το Συμβούλιο γιατί το Συμβούλιο δεν ε, εμπλέκεται επισήμως στο δεύτερο γύρο ε, αυτή η διαδικασία ε, όσον αφορά επίσημους νομικούς όρους δεν εμπλέκει το Συμβούλιο στο δεύτερο γύρο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως παραμένω στη διάθεσή σας. Και τώρα λέει η Πρόεδρος, κυρία Ντελαέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για μία ακόμα φορά που έκοψα το λόγο από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Λοιπόν, σημείωσα προσεκτικά όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων που από ό,τι διαπιστώνω είναι συγκλίνουσες ε, και αυτό αποτελεί καλό ιονό για ε, ικανοποιητική και ε, καρποφόρα συνεργασία. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε ε, να ξεπεράσουμε ε, όλες τις διαδικασίες απόφασης ε, τις οποίες καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε ακόμα και τις πλέον ακαθόδεις και δύσκολες. Και όλα αυτά βεβαίως γιατί θέλουμε να είμαστε στην υπηρεσία των πολιτών και γιατί θέλουμε και οι πολίτες να προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες οι οποίοι αποθαρρύνονται συχνά από την έλλειψη διαφάνειας θα έρθω συντόμως σε επαφή με τους ε, σκιώδεις εισηγητές έτσι ώστε να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα όσον αφορά την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. 18 Ιανουαρίου η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 27 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην ε, ΕΜΒ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το σημείο στη μέρη σε διάταξη. Λοιπόν, όσον αφορά το Λούλουσεφ, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ο επίσημος ε, τριμερής ε, διάλογος. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βρήκαν πολιτική συμφωνία και έχουν καλύψει δι' ε, όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ε, δασοκομεία. Ε, έχει προταθεί από το Συμβούλιο αυξημένη ευελιξία όσον αφορά το θέμα αυτό και συμπεριλαμβάνεται και συμβαστικό κείμενο σχετικά με το πώς θα οριστεί αυτή η ευελιξία. Ορίζεται δε ε, και η περίοδος ε, αναφοράς ε, βάσει της οποίας θα πρέπει να εκδοθούν οι εκτελεστικές, συγγνώμη, οι κα, εξουσιοδότηση πράξης. η διαδικασία αυτή θα γίνει υποχρεωτική για την επόμενη περίοδο εκτός και εάν ε, ε, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας ε, δεν τεθεί σε ισχύ μετά από απόφαση των συνομοθετών. Επίσης, έγινε για το θέμα αυτό τριμερής διάλογος. Να σας πω ότι επιβεβαιώθηκε το, η έκβαση και τα συμπεράσματα των τεχνικών συνεδριάσεων Ε, ε, και υπό την ευελιξία έχουν πλέον συμπεριληφθεί ε, και οι υγροβιότοποι. Οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως τις, τους προσανατολισμούς, τους περιορισμούς, τις τροποποιήσεις κλπ. Έγιναν μακρές συζητήσεις ανοιχνεύτηκαν διάφορες οδοί και εναλλακτικέ λύσεις μέσω και του δομημένου διαλόγου για την Κομισιόν και τους ε, συνομοθέτες έτσι ώστε να προσεγγίσουν οι θέσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά εν τέλει δεν είχαμε συγκεκριμένα ε, αποτελέσματα. Είχαμε και μια πρόταση ε, της Εστονικής Προεδρίας ε, για να ε, ξεκινήσει την 1η Ιουνίου του 2019 η μείωση του μεγέθους της ε, της, ε, του αποθεματικού από 115 σε 105 εκατομμύρια τόνους. Ε, ο εισηγητής ήρθε σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές σε γραφτή διαδικασία λίγο πριν τα Χριστούγεννα και η, η, η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να δεχτεί αυτήν την συμφωνία. Η Κορεπέρ τώρα θα συζητήσει το θέμα αυτό τη 17η Ιανουαρίου, αναμένεται δε να το αποδεχθεί και σε αυτή την περίπτωση η ψηφοφορία στην ΕΜΒΗ θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο στη συνεδρίασή μας στις 24-25. Όσον αφορά τώρα τα απόβλητα στον έκτο ε, άτυπο ε, ανεπίσημο τριμερή ε, διάλογο όσον αφορά την δέσμη για το, για τα απόβλητα, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν συμφώνησαν ε, σε μια τελική ε, συμφωνία προς ώρας για το συνολικό όμως πακέτο ε, που συμπεριλαμβάνει και στόχους και εξαιρέσεις. Κυρίως δε βρέθηκε συμφωνία όσον αφορά τους δεσμευτικούς στόχους για την επανάχρηση και την ανακύκλωση των των κοινοτικών ε, και δημοτικών ε, αποβλήτων, καθώς επίσης ε, και των αποβλήτων συσκευασίας και επίσης οι συνομοθέτες συμφώνησαν ότι θα υπάρξει αναθεωρητική ρήτρα για τους στόχους το 2024. Αυτά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Και με αυτά τα ολίγα και χαρούμενα ολοκληρώθηκε και η ημερήσια διάταξή μας για σήμερα. Όπως σας είπα και στην αρχή της συνεδρίασης, ε, στο Στρασβούργο 15 Ιανουαρίου θα έχουμε μία ε, έκτακτη συνεδρίαση και βεβαίως ισχύει πάντα η συνεδρίασή μας 24